Okay. So, good morning. Good morning, everyone. Καλημέρα. Hmm. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης ε, ως ήθιστε. Έχουμε ανακοινώσεις της Προέδρου και ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους, αλλά αυτό το σημείο θα το εξετάσουμε μετά το σημείο 4. Τώρα θα έχουμε την δημόσια κρόση με τον Αντρέα Ενριεφ εφόσον εγκρίνει τη μερίσια διάταξη, έτσι. Ωραία. Δημόσια κρόση λοιπόν με τον Αντρέα Ενρία. Σας ε, ορίζω ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο του εποπτικού μηχανισμού. Είναι η δεύτερη τακτική ακρόαση που έχουμε με τον κύριο Ενρία εδώ στην Επιτροπή μας το 2019. 4 Σεπτεμβρίου ήταν η προηγούμενη ακρόαση που είχαμε και θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας ε, μεταξύ άλλων και μέτρα ε, για τις τράπεζες το μέλλον της Τραπεζικής Ένωσης και επίσης θέλουμε να θίξουμε μαζί σας και άλλα θέματα, την ε, χρηματοπιστωτική τεχνολογία, την κατάσταση πραγμάτων επίσης της περασκευαστικής εργασίας που έχει γίνει εν του Brexit. Έχετε το λόγο λοιπόν για εισαγωγικες παρατηρησεις παρατηρήσεις, 10-15 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας και πάλι για να συζητήσω μαζί σας το έργο, το εποπτικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις μας για λογοδοσία και διαφάνεια. Συνεχίζουμε πρόοδο για να μειώνουμε τους κινδύνους στο τραπεζικό κλάδο. Η κεφαλαϊκή θέση των τραπεζών υπό τη δικιά μας εποπτεία έχει βελτιωθεί. Επίσης έχει βελτιωθεί και η κατάσταση της μόχλευσης και η ρευστότητα. Ο όγκο τώρα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που διακρατούν οι τράπεζε υπό την δικιά μα άμεση εποπτεία ήταν 562 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ στα τέλη του Ιουνίου του 2019. Όταν ανέλαβε τις εποπτικές αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από 5 χρόνια ήταν 1 τρισεκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγο έχει μειωθεί από το 8% στο 3,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτή τη μείωση διαπιστώνουμε ότι έχει μεταχυθεί τα δύο τελευταία χρόνια και προχώρησα πάρα πολύ γρήγορα σε χώρε που είχαν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο με εξυπηρετούμενων δανείων. Ξεκινήσαμε τη δημοσίευση λοιπόν ε, των κατευθυντήριων γραμμών το Μάρτιο του 2017, κάτι που δείχνει ότι υπήρξε ανταπόκριση. Παρά την πρόοδο όμω σήμερα, το συνολικό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό κλάδο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην ε, αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία των τραπεζών. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε οι προσπάθειες. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την κάλυψη των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συνεργαζόμαστε και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με διάφορες πρωτοβουλίες προκειμένου να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα μη εξυπηρετούμενα ε, δάνεια που διακρατούν λιγότερο σημαντικές ε, τράπεζες. Ο στόχος μας προχωράει. Τα εσωτερικά μας μοντέλα, τα TRIM, σχεδόν ολοκληρώνονται. Υπάρχει εμπιστοσύνη και ο κόσμος θεωρεί ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο σύστημα το οποίο όμως δίνει αποτελέσματα ε, παντού στις τράπεζες. Είναι έλεγχος των εσωτερικών μοντέλων των τραπεζών κατά πόσο μπορούν δηλαδή να μας δώσουν συγκρίσιμα ε, αποτελέσματα. Μετά από τέσσερα χρόνια έχουμε ολοκληρώσει το τελικό στάδιο των ε, ερευνών που κάνουμε on-site των επιθεωρήσεων. Για τις τράπεζες, το TRIM έχει ανεβάσει τον ε, πύχη, προκειμένου να διορθώνει τις διάφορες ελλείψεις. Τα μοντέλα τώρα για, μικρές, για μικρά και πολύ μικρά χαρτοφυλάκια, για παράδειγμα, έχει οδηγήσει σε 20 αποτελέσματα όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων κλειδί. Οι τράπεζες λοιπόν θα βελτιώσουν ε, την ε, κατάστασή τους, τα μοντέλα τους και χρειάζονται βέβαια και νέες προδιαγραφές που τις θέτει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ήδη προχωράει το έργο μας και για τους επόπτες το τρίμη επιβεβαιώνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πόρους για να συνεχιστεί η εποπτεία κυρίως με έρευνες on-site για να διατηρήσουμε υψηλή, υψηλά επίπεδα ποιότητας και προδιαγραφών στο μέλλον. Τώρα, η Βασιλεία 3, εφόσον ε, τεθεί σε εφαρμογή, θα βοηθήσει επίσης ακόμα περισσότερο για τη μείωση του κινδύνου. Θα καλύψει τα κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν καλύφθηκαν από την κρίση. Και είναι βασικό. Η Βασιλεία 3 να υλοποιηθεί πιστά και με συνέπεια και έγκαιρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει τα μαθήματα του παρελθόντος, δεν πρέπει να ξεχάσει τις επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης επί των οικονομιών μας και της κοινωνίας μας γενικότερα. Και επίσης πρέπει να σέβεται και τις δεσμεύσεις της διεθνώς. Οι τράπεζες ε, τώρα ασχολούνται με το τελευταίο στάδιο της Βασιλείας 3. Ε, Αλληνές προδιαγραφές δεν έχουν στόχο μόνο ε, να ανεβάσουν τον πύχη για όλες τις τράπεζες. Έχουν επίσης σαν στόχο τις τράπεζες προκειμένου αυτές να μπορούν να υποφεληθούν καλύτερα από τα εσωτερικά μοντέλα ώστε να υπολογίζουν καλύτερα τις κεφαλικές τους απαιτήσει. Οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές και μια τέτοια αύξηση των κεφαλικών απαιτήσεων είναι αναγκαία. Ένα σημαντικό στοιχείο της, ε, των μεταρρυθμίσεων που έρχονται είναι η εισαγωγή του output floor. Πρόκειται για μια ασφάλεια ώστε τα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών να μην οδηγήσουν ποτέ σε πολύ χαμηλά επίπεδα κεφαλαίων, αλλιώς δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοια μοντέλα οι τράπεζες Και συμπληρώνουν επίσης και το έργο των TRIM. Αποτελεί λοιπόν ένα επίπεδο ασφάλειας για ελεγχιστοποίηση του κινδύνου σε διάφορες ε, τραπεζικές, ε, σε διάφορους τραπεζικούς ομίλους. Για τους διεθνείς μας εταίρους, η μέθοδος αυτή, το output του floor, είναι κάτι το οποίο έχουν ε, συμφωνήσει και αποτελούσε και κόκκινη γραμμή για αυτούς. Όταν κοιτάμε τις επτώσεις της Βασιλείας 3 πρέπει να δούμε και τις ε, κανονιστικές αλλαγές οι οποίες θα οδηγήσουν σε πιο ευθύγραμμες απαιτήσει. Για παράδειγμα, οι κεφαλικές απαιτήσει στην ε, Οδηγία 5 περιλαμβάνουν νέους κανόνες για την ποιότητα του κεφαλαίου και υπάρχει, υπάρχουν και απαιτήσει του πυλώνα 2 που επικεντρώνονται όχι μόνο στο, στη βαθμίδα 1, αλλά και αλλού. Όταν οι αλλαγές αυτές ε, πέρασαν από διαπραγματεύσεις, η εποπτεία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, το είπε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπήρχαν κάποιε ανησυχίε. Σύμφωνα με τους δικού μα υπολογισμού, η αλλαγή θα οδηγήσει σε μία μείωση στι απαιτήσει τη Βαθμίδα 1 σε 90 ε, ε, μονάδες βάσης γιατί θα πρέπει να βασίζονται στα χαμηλά ε, επίπεδα επιπροσθέτως της βαθμίδας 1 και 2. Ως επόπτες μπορούμε να εργαστούμε για να προλάβουμε κάποιες ε, επιπτώσεις της Βασιλείας 3 για τις τράπεζες όσον αφορά τις απαιτήσει του πυλώνα 2. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις στα βάρη που επομίζονται οι τράπεζες. Επίσης, ε, πρέπει να μην κοιτάμε μόνο τις αριθμητικές επιπτώσεις των βαρών από τον πυλώνα 2. Εάν η βασική κίνδυνη συγκέντρωσης ε, καλύπτονται από τον πυλώνα 2, αλλά δεν υπάρχουν αλλαγέ, τότε η αύξηση στι κεφαλαϊκέ απαιτήσει δεν δικαιολογείται. Οι επιπτώσει όμω των νέων προδιαγραφών δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να αντισταθμίζονται πλήρω, γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο του υποπτικού στόχου τη μεταρρύθμισης. Γνωρίζουμε και μα απασχολεί το θέμα τη χαμηλή κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά αν έχουμε χαλαρέ ρυθμίσει και αν ε, παρεκκλίνουμε από τι διεθνεί προδιαγραφέ, αυτό δεν είναι λύση. Αντίθετα, πρέπει να να μείνουν στο επιχειρησιακό τους μοντέλο, να ενισχύσουν τα μέτρα και να υποφελούνται από τις ευκαιρίες που δίνουν νέες τεχνολογίες. Η ψηφιοποίηση θέτει σημαντικές προκλήσεις στις τράπεζες και στους επόπτες οι επιχειρήσεις τέτοιας τεχνολογίας πρέπει να έχουν μια τραπεζική άδεια. Εμείς θα δημοσιεύσουμε κατευθυντήριες γραμμές για να εξηγήσουμε πόσο πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά και πώς τέτοιες εταιρείες FinTech ε, μπορούν να εργάζονται. Και έχουμε και την δημοσίευσή μας για τους κινδύνους και την εποπτεία που λαμβάνουμε υπόψη μας και τον παράγοντα αυτό FinTech και τις επιπτώσεις στις τράπεζες. Επίσης είχαμε και τον πρώτο διάλογο για την χρηματοπιστωτική τεχνολογία και πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τα ρομπότ και το clouding. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να προβλέψουμε πώς η ψηφιοποίηση θα αλλάξει τελικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και τη δομή της αγοράς. Είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερα την ε, ε, προσέγγιση μας στην εποπτεία και να είναι αυτή ουδέτερη. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, ε, έχουμε πρόοδο όσον αφορά τη μίσο των κινδύνων και τις ε, ρυθμίσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την γενική αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης. Η, τα πλαίσια διαχείρισης της κρίσης πρέπει να βελτιωθούν, διότι παραμένει κατακαιρματισμό και κάποια εργαλεία λείπουν ακόμα ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο για την έγκαιρη ε, παρέμβαση πρέπει να αναθεωρηθεί για να απλοποιηθούν οι κανόνες και να διευκρινιστεί και η σχέση μας με άλλα εποπτικά μέσα. Επίσης κάποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, μαθαίνοντας από άλλες ε, νομολογίες. Το θέμα της εξυγίανσης, για παράδειγμα, είναι κάτι που εφαρμόζεται με 19 διαφορετικές εθνικές διαδικασίες. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες για να ξεκινάνε οι διαδικασίες εξυγίανσης, πώς ε, γίνεται η ταξινόμηση και τα εργαλεία ακριβώ που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Χρειαζόμαστε πραγματικά διαδικασίες ε, εκαθάρισης που να είναι ομοιόμορφες για τις τράπεζες. Μπορούμε να μάθουμε φυσικά από τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, με τις νέες διοικητικές εξουσίες που αναλαμβάνει ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίασης. Έπειτα έχουμε και το έντις που είναι ο τρίτος ο πυλώνας, εγγύηση καταθέσεων δηλαδή που δεν ε, υπάρχει ακόμα. Ε, χρειάζεται για να εκτεθεί εμπιστοσύνη των καταθετών και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλες τις χώρες μέλη. Επιπλέον, έτσι δεν θα χρειάζεται άλλη δικαιολογία για τους κανόνες και τις πολιτικές που απαιτούν την πλήρη ολοκλήρωση γιατί θα έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά από την Τραπεζική Ένωση. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνεχιστεί και να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για την νομισματική και τραπεζική ένωση. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφερθώ και στο Brexit. Εμείς ε, τονίζουμε ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες λειτουργικά όσο γίνεται πιο γρήγορα και συνεχίζουμε να προοδεύουμε όσον αφορά την εφαρμογή των μοντέλων λειτουργίας τους που έχουμε αποφασίσει σύμφωνα με τα προηγούμενα χρονοδιαγράμματα έτσι όπως είχαν αποφασιστεί εν ώψη του 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ενρία. Αρχίζουμε ε, σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Η κυρία Περέιρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Καλώς ορίσατε κύριε Εριά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις που είναι περίπλοκες, ε, ποικίλε ε, και πάρα πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη θα πρέπει με ένα ομαλό και γρήγορο τρόπο να, να δούμε πώς θα αυξηθεί η ανάπτυξη. 1,1% αναμένεται για το 2019 ε, που ε, σύμφωνα με τις περισσότερες προβλέψεις υπολείπεται κατά 0,7% και δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Οι οικονομίε μας λοιπόν έχουν διάφορες προκλήσεις για την κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση κτλ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση. Αυτή μπορεί να έρθει μόνο από μεγαλύτερη ανάπτυξη και πιο βιώσιμη. Ο τραπεζικός τομέας έχει εδώ να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μεταρρυθμίσαμε σε όλη την Ευρώπη μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του τραπεζικού τομέα, αλλά απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Και θα πρέπει επιγόντω να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, όπω είπατε, με τον τρίτο πυλώνα, για παράδειγμα. Αλλά σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup ε, δεν βγάζουν συμπεράσματα για το ίδις. Ε, θα πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εκαθάριση και εξυγίαση και κάποιες τράπεζες ε, που είναι ακόμα ε, σε προβληματική κατάσταση. Ξέρουμε ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης ε, δρούν σε ένα περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια και αυτό είναι ο κίνδυνος για τους στόχους κερδοφορίας τους. Και επίσης, έχουν και κάποιες τράπεζες που έχουν συγχωνευτεί στην εξυγίανση ε, και δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο. Το αντίστοιχο ταμείο ε, έχει κληθεί να δώσει από το 2014 πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η εξυγίαση μπορεί να στηρίξει τις τράπεζες και το δημόσιο αυτό χρήμα να επανεπενδύεται σε παραγωγικές επενδύσεις για την οικονομία. Είπατε ότι υπάρχουν διάφορα πλαίσια, 26 τον αριθμό, διαφορετικά εθνικά. Πώς όμως θα οδηγηθούμε σε πιο παραγωγικές και πιο επιτυχείς ε, λειτουργούσες τράπεζες, αφού έχουν περάσει από όλους αυτούς τους και καιρούς. Ευχαριστώ απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Έχετε δίκιο. Αν κοιτάξετε τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε με την κληρονομιά της κρίσης είναι ότι είναι πολύ λίγη ε, η ε, αναδιάρθρωση των τραπεζών και έγινε και πάρα πολύ αργά θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να επιτρέπει εγκαίρως νωρίς να επεμβαίνουμε στις τράπεζες και να τις πιέσουμε να μπουν σε μια διαδικασία ε, για να μπορέσουν να ε, ε, στηρίξουν την οικονομία όσες τράπεζες επιβιώσουν. Και αν δούμε τι έγινε με τις προσαρμογές στις ευρωπαϊκές και στις αμερικανικές τράπεζες, οι Αμερικανοί αντέδρασαν πολύ πιο γρήγορα και καθάρισαν τους ισολογισμούς, επανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες και μείωσαν τον αριθμό των τραπεζών. 500 τράπεζες ε, στα τρία χρόνια μετά την κρίση βγήκαν από την αγορά. Αυτό δείχνει λοιπόν ε, ότι οι τράπεζες έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία και μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα την οικονομία. Ε, στην Ευρώπη δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το είδος του συστήματος και είμαστε πιο αργοί. Έχουμε κάνει πρόοδο για να είμαι ειλικρινής και ε, αναδιαρθρώθηκαν οι τράπεζες νομίζω θετικά για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την κληρονομία των τραπεζών, να καθαρίσουμε τους ισολογισμούς τους, να απλοποιήσουμε τις δομές για να μπορέσουν και πάλι οι τράπεζες να στηρίζουν την οικονομία. Και βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο δανεισμός τα τελευταία χρόνια ε, χορηγήσεις που δείχνουν ότι λειτουργεί καλύτερα ο ευρωπαϊκός τραπεζικός ε, κλάδος. Πάντως ε, θα έλεγα ότι δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι και η πραγματική πρόκληση θα είναι αυτή η ταχύτητα. Και όπως είπα και προηγουμένως, ε, αναφέρθηκα στο FDIC που είναι το αμερικανικό σύστημα. Εκεί υπάρχει μια αρμόδια αρχή η οποία αναλαμβάνει τις τράπεζες που πτωχεύουν ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν και μεταφέρουν το ενεργητικό και το παθητικό των τραπεζών αυτών σε άλλες τράπεζες, κυρίως από άλλες πολιτείες έτσι συνήθως και αυτό βοηθάει και όλα το γενικό σύστημα στην Αμερική. Ε, χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα διοικητικό εργαλείο για την εκαθάριση των τραπεζών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσουμε στους επιθυμητούς στόχους. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταστάσεις όπου οι τράπεζες ε, ε, κηρύσσονται σε πτώχευση ότι κινδυνεύουν, τις χαρακτηρίζουμε έτσι, δεν περνάνε τα, τις ε, δοκιμές, δεν μπαίνουν στην εξυγίαση από το αντίστοιχο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εθνικό πτωχευτικό δίκαιο δεν θεωρούνται υποπτώκευση και παραμένουν εκεί μετέωρες για κάποια χρόνια, ε, έχουν άδεια να λειτουργούν ως τράπεζες, ε, αλλά ε, είναι μια κατάσταση προβληματική. Θα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή λύση για αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χώνας Φερνάντεθ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίσατε. Καταρχάς, συμφωνώ κύριε Ρία μαζί σας στην περιγραφή που κάνατε της Τραπεζικής Ένωσης για τα προβλήματα συνοχής που υπάρχουν και συνέπειες. Ακούτε? Αλλά μην ανησυχείτε. Sí. No, le decía Λέγα ότι συμφωνώ στην περιγραφή που κάνατε της σημερινής κατάστασης και στα προβλήματα συνοχής και συνέπειας που έχουμε ε, στο σχεδιασμό ε, της σημερινή Τραπεζικής Ένωσης. Το, το ε, δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί και δεν μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα εξυγίανσης και καθάρισης των τραπεζών με κάποια συνέπεια. Και τώρα, αν πρέπει να εναρμονιστεί ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η πτώχευση των τραπεζών. Αλλά τι γίνεται με την έμεση εποπτεία ε, κάποιων οργάνων στην Τραπεζική Ένωση. Εκεί δεν εμφανίζονται προβλήματα συνέπειας. Βλέπουμε και κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις για να σωθούν κάποιες τράπεζες. Μιλώ για τη γερμανική περίπτωση. Αυτή η έμεση λοιπόν εποπτεία κάποιων τραπεζών και κάποιων οργάνων που εσείς έχετε υπό την άμεση εποπτεία σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες ε, ασυνέπειες στο μοντέλο αυτό. Και μια δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει περισσότερο με τα βιώσιμα οικονομικά. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χτες κατέθεσε ένα πρόγραμμα για να πλαισιώσει αυτό το έργο τα επόμενα χρόνια και μάλλον το τελευταίο τρίμηνο του 2020 θα φέρει μια πρόταση για τα βιώσιμα οικονομικά όπου σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει ε, διαφορετικές ε, κεφαλαιακές απαιτήσει για ε, αυτά στις, τα πράσινα δάνεια. Εσείς ως επόπτης πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ για το πρώτο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν στην περίπτωση του Northern Bay, που είναι υπό άμεση εποπτεία της ΕΚΤΑ και είναι ένα σημαντικό πιστοτικό ίδρυμα. Τα πρόβλημα συνέπειας που βλέπουμε σε αυτόν τον τομέα, βεβαίως για λιγότερα σημαντικά ιδρύματα, έχουμε παρακολούθηση και εποπτεία των δράσεων των εθνικών αρχών. Οποτεδήποτε υπάρχει μια τράπεζα που είναι κοντά σε κρίση, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και αρχίζουμε τις εργασίε και συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές αρχές. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορέ έχουμε διαφορετικές νομοθεσίες ε, και διαφορετικές δομές σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να αλληλεπιδράσουν διαφορετικά όταν υπάρχει κρίση. Αυτό ακριβώ ανέφερα προηγουμένω. Ανέφερα την καθάριση και του κανόνε καθάριση και εξυγίανση. Το ίδιο όμω ισχύει για τους κανόνες ε, για το σχήμα μετά τις εγγύησεις. Όταν θέλουμε να κάνουμε αναδιάρθρωση σε περίπτωση κρίσης. Αυτό έγινε στην Ιταλία. Με την παρέμβαση του υποχρεωτικού και θελωτικού τμήματος του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Και στην Γερμανία, στην περίπτωση του Northern Bay, έχουμε ε, ένα μεικτό σύστημα θεσμικής και μη προστασίας που παρενέβη και τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να παρέμβει το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τελείως διαφορετικά από κράτο μέλλον. Μερικές φορές παρεμβαίνει προληπτικά εφόσον δεν υπάρχει κάποιο στην νομοθεσία, ενώ μερικές φορές είναι τελείως απόλυτα εκτεταμένη η παρέμβαση. Θα πρέπει να υποφεληθούμε από αυτές τις δυνατότητε λοιπόν και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη Μπάνκα Τέρκας για να υπάρξει μια πιο ομοιόμορφη ε, παρέμβαση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων σε περίπτωση κρίσης και να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτό το κομμάτι για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση η θέση μου ήταν πάντα ότι οι προνοιακές ε, ε, προϋποθέσεις, θα πρέπει να συνάθουμε τον κίνδυνο. Αν υπάρχει ένα τομέας ε, δραστηριότητας λιγότερο επικίνδυνος, θα πρέπει να έχει λιγότερο κεφαλιακές απαιτήσει και αν είναι περισσότερο επικίνδυνος, θα πρέπει να έχει περισσότερες. Επίσης, για την πράσινη χρηματοδότηση μερικές φορές θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την χορήγηση λιγότερου κεφαλαίου. Ε, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε καλά τι σημαίνει οι κεφαλιακές ε, απαιτήσεις. Θεωρούμε ότι αυτό, αυτή η χρηματοδότηση ε, αφορά την οικονομία. Αλλά στην πραγματικότητα ε, χρηματοδοτούνται οι τράπεζες έτσι. Και όσο καλύτερα χρηματοδοτούνται μπορούν να, να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους και να υποστηρίξουν καινοτόμα τμήματα της οικονομίας. Εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε ε, την μετάβαση από την ε, καφέ ας πούμε στην πράσινη οικονομία υπάρχουν ε, κανόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Όταν χρησιμοποι... Ε, συζητήσαμε τις ε, προληπτικές απαιτήσει ή όταν τη συζητάμε, θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Thank you. Συνεχίζω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ο κύριος ε, Γκαρικάνου. Μας εξέπληξε η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για να μην διασωθεί η Northern Bay. Σε άλλες περιπτώσεις έγινε μια μεγάλη κρατική παρέμβαση, 4,8 δισεκατομμύρια έγχυση κεφαλαίου. Στη Northern Bay έχουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,3 εγγύηση των περιουσιακών στοιχείων ε, από φορολογούμενους, 1,3 δις. Ε, χρησιμοποιούμε δημόσια κονδύλια για να διασώσουμε αυτές τις τράπεζες. Μήπως το σύστημα εξυγίανσης δεν είναι αρκετά αξιόπιστο. Ε, μερικές φορές ε, είναι καλύτερα να καθαρίσουμε με εθνικούς κανόνες αυτές τις τράπεζες. Ε, δηλαδή υπό την έννοια ότι καλύτερα να τις αφήσουμε να πεθάνουμε, να πεθάνουνε γιατί τώρα τις, τις στάβουμε σε χρυσά, ας πούμε, φέρετρα. Εσείς πιστεύετε ότι η Northern Bay έχει αντιμετωπίσει, την έχουμε αντιμετωπίσει σωστά και κάτι που μας ενδιαφέρει για τράπεζες ζόμπι, ε, νεκροζώντανες. Ε, λειτουργούν, ας πούμε, έχουν την τραπεζική άδεια, αλλά δεν λειτουργούν ουσιαστικά. Η πρόεδρος της SRB ανέφερε πρόσφατα το εξής, ότι θα, θα μπορούσε ε, σε αυτή την περίπτωση να επιτρέπουμε στην, ε, στο σύστημα, στο SSM, να αποσύρουν, να αφαιρούν την άδεια των τραπεζών. Μήπως ήταν αυτή μια καλή λύση. Θα το να κρατούν ακόμα την άδεια και ουσιαστικά να υπολειτουργούν. Δύσκολο ερώτημα, λέει ο κ. Σενρία. Φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ εξ ονόματος της ε, Κομισιόν για το θέμα των ε, κρατικών ενισχύσεων, αλλά συνεργαζόμαστε μαζί. Κοιτάμε ε, την, την υπόθεση από εποπτική άποψη. Τι προβλέπει η νομοθεσία, επίσης κοιτάμε. Ειδικά με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, για να αξιολογήσουμε το κεφαλαιακό και επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας. Αν είναι βιώσιμο από προληπτική σκοπιά, αν η τράπεζα θα μπορούσε βιώσιμα να σεβαστεί τις κεφαλαιακές απαιτήσει και οι συνάδελφοι στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού κοιτάνε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Η αξιολόγηση του σχεδίου των τραπεζών γίνεται συντονισμένα με την Κομισιόν. Κατάλαβα επίσης και την ε, αντίληψη ότι το πλαίσιο εξυγίανσης μπορεί να μοιάζει ανεπαρκές, ατελές. Καταρχάς αυτός που, αυτό που αναφέρατε σωστά, ότι η κρέδιτος μπορεί να εκαθαριστεί καλύτερα σε εθνικό επίπεδο παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. δεν θα πρέπει κατά την εκαθάριση, ας πούμε, κάποιοι πιστωτέ να βγαίνουν κερδισμένοι και κάποιοι όχι. Αυτό το ανέφερα προηγουμένω. χρειαζόμαστε πιο εναρμονισμένο πλαίσιο για την ε, εκαθάριση. Επίσης, υπάρχουν ε, πρωτοβουλίε για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διαδικασιών ε, πτώχευση Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια διοικητική εκαθάριση εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση δημοσίων κονδυλίων. Η περίπτωση της Northern Bay είναι μια τράπεζα δημόσια. Όταν η τράπεζα δεν σέβεται τις ε, προϋποθέσεις, τότε ο επόπτης ζητάει από την τράπεζα να φτιάξει ένα σχέδιο για να συμμορφωθεί εκ νέου με τις προϋποθέσεις. Και γενικά η τράπεζα πάει στους ε, μετόχους για να τους ε, ζητήσει κεφάλαιο, ούτω ώστε να μπορέσει να υπάρξει συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Αυτό συνέβη σε αυτήν την περίπτωση και αυτό που είναι κρίσιμο είναι οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες που η Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θέτει, ε, ούτως ώστε το σχέδιο αυτό να συμμορφούνται με την αγορά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Συνολικά νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε είναι συχνά έχουμε τις τράπεζες που σέβονται τις προϋποθέσεις αλλά έχουν επιχειρηματικό μοντέλο που δεν είναι βιώσιμο. Είναι ένα τομέα παρέμβασης για εμάς τις εποπτικές αρχές που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Φυσικά, ζητάμε από τις τράπεζες να παρέμβουν και να διορθώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, όπως, έχουμε, όπως στην περίπτωση της της Κάισα, ε, τα μέτρα μας είναι πολύ πανεβατικά, αλλά δεν μπορούμε συχνά, ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια αυτό και δεν μπορούμε να υποκαθιστούμε το, τη διοίκηση της τράπεζας όταν δεν σέβεται τις προϋποθέσεις. Ε, το να αποσύρουμε την ε, άδεια της τράπεζας είναι ακραίο μέτρο που έρχεται μετά τη διαδικασία φερεγκαιότητας της τράπεζας. Το να παρέμβουμε, παραδείγματος χάρη στην ε, Anglo-Austrian Bank, όπου οι υποπτικές αρχές της Αυστρίας δεν πήραν απόφαση και έχουμε, μία, έχουμε μπει σε μια διαδικασία αφαίρεσης της άδειας, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σταμάτησε αυτή τη διαδικασία. Ελέγχουν τι άλλε ε, δυνατότητες υπάρχουν και μόνο όταν δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα τότε αφαίρουμε την άδεια της τράπεζας. Είναι πολύ περίπλοκο λοιπόν το θέμα. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκικόλτ τώρα. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στη Λαβαλέτα, στη Μάλτα. Και επί τη ευκαιρία αυτή Είδα και την έκθεση Reuters για την αδυναμία της τράπεζας της Βαλέτα, μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες εκεί. Και διάβασα και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να σχολιάσετε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ήταν μια καταδικαστική έκθεση και ευχαριστώ που τα παρακολουθείτε, αλλά πραγματικά με σοκάρει εμένα που μπορεί να φτάσουμε σε μια τέτοια εξέλιξη ε, με μια τράπεζα που βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Συνεπώς, μία ερώτηση έχω. Έχετε την υποχρέωση να κάνετε σωστή αξιολόγηση σε όσους βρίσκονται σε ηγετική θέση στις τράπεζες. Μπορείτε να μας πείτε πόσο συχνά ο SSM ή το έκανε ποτέ να πει όχι για οποιονδήποτε από τότε που δημιουργήθηκε ο μηχανισμός αυτός, ο εποπτικός. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τα στατιστικά στοιχεία μαζί μου, αλλά για να λέμε την αλήθεια δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ σημασία, γιατί συμβαίνει συχνά ε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται να τίθονται επεξέταση και τελικά η τράπεζα να μην συνεχίζει με τον ορισμό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Δεν έχω τα στατιστικά δεδομένα, αλλά να ξέρετε ότι συμβαίνει αρκετά συχνά. Τώρα αυτό που θέλω να σας πω είναι για ένα νέο εργαλείο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η ιδέα αυτή του fit and proper, της καταλληλότητας δηλαδή, δεν είναι μια εκτίμηση που γίνεται μια και έξω δηλαδή όταν ε, κάποιος ε, πάει ορισμό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σε συνεχή βάση. Δηλαδή να αναθεωρούμε και όλα κατά πόσο κάποιος είναι κατάλληλος βάσει νέων στοιχείων. Και όταν υπάρχουν περίπτωση κακής διαγωγής για παράδειγμα ή κακής απόδοσης ε, στο θέμα του, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομα χρήματα ή εσωτερικών ελέγχων κλπ εμείς έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιούμε περισσότερες ε, εκθέσεις, να ψάχνουμε να βρούμε ποιο μέλος ήταν υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες λειτουργίες και ποιος είναι αυτός που τελικά δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια καταλληλότητας. Και συνεχίζεται η προσπάθεια. Μπορώ να κάνω συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ωραία. Σε μία ομιλία, μάλλον να το πω αλλιώς. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις και οι δυσκολίες. Ναι, αλλά πόσο ξέρω εγώ, ποτέ δεν συνέβη ο SSM να πει όχι σε κάποιον υποψήφιο. Ε, ναι, κάνετε δύσκολες ερωτήσεις, σύμφωνοι, αλλά δεν λέτε ποτέ όχι. Οπότε, καλό θα ήταν να είχαμε τα νούμερα. Πόσους υποψηφίους έχετε γκρίνει πώς, σε πόσους υποψήφιους είπατε όχι και για πόσους υποψηφίους γνωρίζετε ότι αποσυρθήκαν τελικά μετά από τις δικές σας ερωτήσεις. Θα βοηθούσαν είχαμε αυτά τα στοιχεία. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι που έχει να κάνει με κάτι που είπε τον Ιανουάριο του 2016 η Σαμπίνε Λάντοσνιτο που μίλησε για την έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά την ε, νομική ρύθμιση της καταλληλότητας. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, έχετε δίκιο. Οι προκλήσεις που βάζετε ε, έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά αν δεν λέτε και όχι σε κανέναν, Μήπως αυτό οφείλεται στην έλλειψη εναρμόνισης. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι θα επιθυμούσατε εσείς να εναρμονίσουμε εμείς για να μπορείτε να κάνετε εσείς καλύτερα τη δουλειά σας. Όντω, ναι, το ξέχασα αυτό το σημείο στην απάντησή μου, λέει ο κύριο Ενδρία, και τώρα θα το κάνω. Ναι, ναι, πράγματι είναι πολύ σημαντικό για μα, γιατί ε, βλέπετε, εμεί έχουμε 19 διαφορετικού τρόπου για να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις και φυσικά δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε αν είναι κατάλληλος κάποιος ή δεν είναι. Αν πρόκειται για τράπεζες σε διαφορετικές χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και έχουμε μια πολύ διαφορετική εφαρμογή λοιπόν και όντως υπάρχουν περιπτώσεις όπως στην Ιταλία όπου η οδηγία δεν εφαρμόστηκε πλήρως η τέταρτη. Όντω είναι πολύ δύσκολο για μα να εφαρμόζουμε τα ίδια εργαλεία με τον ίδιο τρόπο παντού. Οπότε η απάντηση είναι απλή. Ναι, να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη εναρμόνιση και τα κριτήρια αυτά να είναι σε κανονισμό και όχι σε οδηγία. Στην Τραπεζική Ένωση πρέπει να έχουμε τα ίδια κριτήρια για όλου. Τώρα για τα στατιστικά δεδομένα, να διευκρινίσω ότι σε πολλέ περιπτώσει, στι περισσότερε μάλιστα, εγκρίνουμε τους ορισμούς υπό όρους, υπό προϋποθέσεις. Αν δηλαδή βρούμε κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης ή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να αφιερώσει το άτομο στις αρμοδιότητές του, ε, τότε βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις. Και φροντίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν από κάποια κατάρτιση για να καταστούν κατάλληλοι. Παρακαλώ να μας στείλετε τα στατιστικά στοιχεία, λέει ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιουτζίνι Αρζίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, οι σημαντικές τράπεζες έχουν χάσει κατά μεσόωρο την κερδοφορία τους. Η ΕΚΤ, εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει μελετήσει λεπτομερώς τις αρνητικές παρενέργειες της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της. Ε, μία από αυτές μπορεί να είναι ακριβώς η χαμηλή κερδοφορία του τραπεζικού τομέα και μπορεί να επιδεινωθεί με το χρόνο. Ερωτώ, εσείς θα πιέσετε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αξιολογεί τεκτικά και να λέει ε, ποιες είναι οι παρενέργειες αυτής της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής. Εδώ στο, το Μάρτιο του 19 στην Επιτροπή μας δεσμευτήκατε να προχωρήσετε σε εποπτικά μέτρα ε, σε τράπεζες που έχουν έκθεση σε δημόσιο χρέος. Πρόσφατα αυξήθηκε αυτό ε, σε σχέση με κάποια αμφιλεγόμενα κρατικά ομόλογα. Ποια είναι τα μέτρα λοιπόν που έχετε λάβει για να ε, καταπολεμήσετε αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για την ερώτησή σας. Για τη χαμηλή κερδοφορία είναι γεγονός ε, ότι είναι χαμηλά τα επιτόκια και αυτό πιέζει τα περιθώρια των τραπεζών. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αν θέλετε όμως να αξιολογήσετε ε, κατάλληλα και σωστά τον όλο αντίκτυπο, θα πρέπει να δούμε και ε, τον παράγοντα της κάθε χώρας. Τα χαμηλά επιτόκια ευνοούν την αύξηση ε, του δανεισμού και τα συνολικά ποσά και φυσικά υποστηρίζουν και την δυνατότητα των δανειζομένων να εξοφλούν τα δάνειά τους και βελτιώνεται και η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Και αν δεν υπήρχε αυτή η ποσοτική χαλάρωση, δεν θα μπορούσαν ενδεχομένω οι τράπεζε να επιτύχουν την πρόοδο που έχουν εμφανίσει τα τελευταία χρόνια στη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ε, κόκκινων δανείων. Είναι γεγονό ότι επηρεάζεται όντω η κερδοφορία των τραπεζών και φαίνεται αυτό πια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι συνάδελφοί μου στη νομισματική πολιτική αναλύουν σε βάθος. Έχουν δημοσιευθεί και αντίστοιχα έγγραφα και αναλύσεις για αυτό το θέμα. αναγνωρίζουμε αυτές τις παρενέργειες και αυτό φάνηκε από τα πρόσφατα μέτρα σε σχέση με την ε, ταξινόμηση, κατάταξη των αποθεματικών ε, στις κεντρικές τράπεζες σε σχέση με τα επιτόκια. Για τις τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε δημόσιο χρέος, με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο, μελετούμε αυτό το κίνδυνο στο πλαίσιο του πυλώνα 2, ας πούμε στις δοκιμές αντοχής στα stress test που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή κάθε δύο χρόνια και το 2020 θα φέρουν καινούργια ε, πρόταση. Αυτό αφορά λοιπόν την έκθεση και τη διασπορά ε, στο δημόσιο χρέος και στην ε, θέση την κεφαλιακή και την έκθεση των τραπεζών. Φυσικά στο δεύτερο πυλώνα μπορούμε να δούμε και με ποιο τρόπο οι τράπεζες ε, παρακολουθούν αυτό το συγκεκριμένο ρίσκο. Υπάρχει κίνδυνο συγκέντρωσης επίσης ε, σε τράπεζες που έχουν κρατικά ομόλογα. Αυτό το παρακολουθούμε τακτικά και όταν εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα δάζουμε και ειδικέ απαιτήσει στις τράπεζες. Κάτι που είχα πει στο παρελθόν και θα ήθελα να επαναλάβω είναι ότι από την παρελθούσα εμπειρία μου στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δίνεται πολύ μικρή προσοχή στη λογιστική διαχείριση του δημοσίου χρέους. Έχουν αυτή την πρακτική που δεν μου αρέσει καθόλου οι τράπεζες να μεταθέτουν τον κίνδυνο ε, ε ε, από τα λογιστικά βιβλία της εμπορικής διαχείρισης ε, ε, στα άλλα βιβλία, τα κεντρικά της τράπεζας, και αυτό δεν επιτρέπει ε, την ε, σωστή ε, αναγνώριση και ανείχνευση των απολειών που έχουν από κρατικά ομόλογα και δημόσιο χρέος. Και έχουν υποχρέωση ρευστότητας οι τράπεζες και όταν υπάρχει σοκ ρευστότητας θα πρέπει πολύ γρήγορα να τα ρευστοποιούν αυτά οι τράπεζες για να ανταποκρίνονται στις κεφαλαϊκές τους απαιτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Χωσέ Γκουσμάου. Κύριε Ανδρία, θέλω να επανέλθω σε κάτι που είπατε. Για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τα λεγόμενα πράσινα περιουσιακά στοιχεία. Άκουσα ήδη τις απαντήσεις σας σε αυτή την ιδέα. Και άκουσα και αυτά που είπε ο κύριος Ντομπρόφσκης, που είπε ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο σοβαρά αυτή την ιδέα. Νομίζω όμως ότι τα επιχειρήματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα επιχειρήματα που πρότεινε είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, ότι το να κάνουμε την τραπεζική δραστηριότητα πιο επικίνδυνη δεν είναι σωστός τρόπος για να προωθήσουμε τις πράσινες επενδύσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά πράσινες επενδύσεις. Τα επιχειρήματα όμως που χρησιμοποίησατε είναι σωστά. Δεν μπορούμε να ζητούμε υψηλότερες κεφαλιακές απαιτήσει για δραστηριότητες που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Όταν λέτε ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσει θα πρέπει να παίζουν το ρόλο τους, παρά να τις χρησιμοποιούμε για διαφορετικούς στόχους, τι πιστεύετε για αυτό που σας είπα πριν, για τις ρηπογόνες δραστηριότητε, ας πούμε, και τις σχέσεις με τις κεφαλαιακές απαιτήσει. Επίσης, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Είναι απαιτήσεις προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Χρειαζόμαστε επιμερισμό των ευθυνών. Πιστεύετε ότι ο στόχος που θέτεται, ότι όλες οι χώρες πρέπει να προστατεύονται εξίσου σε ό,τι αφορά το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή μέσω αυτού του συστήματος, θα μπορούσε να συμπληρωθεί με ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων που βασίζεται στον δανεισμό. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σας σημείο, να σας πω αμέσως ότι ο επίτροπο ζήτησε από την EBA, από την Εποπτική Αρχή των Τραπεζών, να κάνει μια ανάλυση και η εποπτική, Τραπεζική Εποπτική Αρχή το εξετάζει. Και συνεισφέρει ούτω ή και θα συνεισφέρει σε αυτή τη δουλειά. Ε, θα γίνει λοιπόν μια ανάλυση. Αυτή η συζήτηση, όπως είπα και προηγουμένω, πρέπει να βασιστεί σε εμπειρικά στοιχεία. Υπάρχει κίνδυνος Υπάρχει μάλλον στοιχεία ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες από ό,τι σε σχέση με κάποιες άλλες. Σε ό,τι αφορά ε, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έγινε μία ανάλυση ε, ότι όταν έχουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι λιγότερο επικίνδυνο από το να έχουμε μονομερή έκθεση σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδίου μεγέθους και αυτό μειώνει ε, και την ε, κεφαλαιακή απέτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, εξάλλου και αυτό αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της Βασιλείας. Τέτοιου τύπου εμπειρική ανάλυση χρειάζεται να κάνουμε. Αυτό που είπατε επίσης είναι σωστό. Εάν θέλουμε να περάσουμε από την πράσινη, στην, από την μπλε, συγγνώμη, την καφέ στην πράσινη οικονομία, κάποιες δραστηριότητες είναι πιο επικίνδυνες και κάποιες άλλες, και κάποιες λιγότερο. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την ε, βιωσιμότητα. Οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το πράγμα μακροπρόθεσμα. Δηλαδή να εξετάσουν τους μακροπρόθεσμους κινδύνους. Τώρα ε, εξετάζουμε τα εσωτερικά μοντέλα και την εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου. Ε, τώρα έχουμε έναν ορίζοντα, ας πούμε, ένα χρόνο ή σε κάποιες τράπεζες τρία χρόνια. Το, να πιέσουμε τις τράπεζες να δουν τον, τον κίνδυνο μέσα σε ένα μακρό πρόθεσμο ορίζοντα και να δούμε ποιες παράμετροι γίνονται πιο σημαντικές ε, επειδή ο ορίζοντας μακραίνει, ε, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ε, εποπτική διαδικασία. Και αν θέλουμε, ας πούμε, να πούμε ποιε είναι οι προσδοκίε μα ό,τι αφορά τα προληπτικά θέματα στι τράπεζε, θα πρέπει αυτού του κινδύνου και τη διαφοροποίησή του όταν έχουμε ακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα να τι λάβουμε υπόψη μα. Τώρα, αν έχουμε ένα μόνο παράγοντα για το, τις πράσινες δραστηριότητες ε, και είναι θετικό και αρνητικός για τα, τις καφέ δραστηριότητες, δεν νομίζω ότι είναι αρκετή διαφοροποίηση. Τώρα, για την για το δανεισμό. Θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση των πόρων και διαφοροποίηση του κινδύνου και για το κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Το ίδιο ακριβώς ποσό, το οποίο προστατεύει τους καταθέτες. Μερικές φορές κάτι που ξεχνάμε στη συζήτηση είναι ότι αυτά τα ε, κονδύλια τα πληρώνουν οι τράπεζες. Ακόμα και αν υπάρχει στήριξη από το κράτος, σε, σε περίπτωση που το σύστημα εγγύης των καταθέσεων δεν μπορεί να ε, τις υποστήριξει, τελικά θα συνεισφέρουν εκ των υστέρων οι τράπεζες και με ιδιωτικά κονδύλια για να υπάρξει μια αντιστάθμιση. Πάντως το να ξεκινήσουμε με δανεισμό, ας πούμε, η στήριξη της ρευστότητα, αυτό είναι μια καλή ε, ιδέα. Επίσης, ε, ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η αντασφάλιση. Και αυτό είναι ένα βήμα ότι κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε, κύριο Μαρτισέλο. Ευχαριστώ. Τρεις ε, σύντομες ερωτήσεις. Χθε το Ιταλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτό το ψήφισμα που εξαρτά την έγκριση της ε, σύνθεσης της ε, συνθήκης του μηχανισμού σταθερότητας από ένα πακέτο με κανόνες για την ε, Τραπεζική Ένωση. Και μιλάει για μια γενική εγγύηση των καταθέσεων. Τι αξία έχει κατά τη γνώμη σε αυτό το ψήφισμα. Δεν θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει φόβους στους οικονομικούς φορείς και δεν μπορεί να δημιουργηθεί πεποίθηση ότι η Ιταλία είναι μια χώρα που χρωστάει. Επίσης, πρόσφατα είπατε ότι για να υπάρξει ενοποίηση στον τομέα, η εποπτεία δεν θα απαιτεί επιπλέον κεφάλαια σε περίπτωση συγκεντρώσεων. Αλλάζει η τάση για την εποπτεία των τραπεζών. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλάζει στάση απέναντι της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τράπεζα, στάση απέναντι ε, κεντρικές τράπεζες. Επίσης η Λαϊκή Τράπεζα του Μπάρι ζήτησε ένα διατραπεζικό δάνειο για τη διάσωσή της. Ε, μέσω αυτού του σχεδίου όμως θα υπάρξει άμεση εμπλοκή του κράτους. Μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ε, αυτό μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση κατά την απόψή σας, αυτό το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Θα αρχίσω από τα εύκολα, που είναι η τελευταία σας ερώτηση. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να αποφασίσουμε για την κρατική ενίσχυση, οπότε δεν θα ήταν σωστό εγώ εδώ να εκφράσω γνώμη από πλευράς κρατικής ενίσχυσης ή όχι. Η τράπεζα της, του Μπάρι σίγουρα είναι λιγότερο σημαντική τράπεζα υπό εποπτεία από την τράπεζα της Ιταλίας αλλά βεβαίω και είμαστε σε επαφή με τις ταλικές αρχές για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM, Ανησυχώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Όταν συζητάει κανείς με χώρες μέλη, ποτέ τελικά δεν έχει μια τελική συμφωνία. Ε, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στο τέλος της διαδικασίας ε, για το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων και ξέρω ότι είναι ευαίσθητα ζητήματα αυτά και λεπτά γιατί έχει να κάνει και με την ε, έκθεση σε δημόσιο χρέος αλλά κανονικά πρέπει να έχουμε χαρτοφυλάκια στις τράπεζες περισσότερο διαφοροποιημένα. Να μην είναι όλες οι τράπεζες με χαρτοφυλάκια από το Ιταλικό χρέος και όλες οι γερμανικές τράπεζες με χαρτοφυλάκια από το Γερμανικό χρέος και το καθεξής. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή ώστε η διαδικασία να προχωρήσει τις διαφοροποίησεις. Και όσον αφορά την άποψη των τραπεζών, που είναι δικιά μου αρμοδιότητα, τι έκανε ο ESM, εφρόντισε να υπάρχει μια προστασία με το Ταμείο Εξυγίανσης. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει να έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διαχειρίζεται την έξοδο από την αγορά, ακόμα και σε περίπτωση μεγάλων και περίπλοκων τραπεζών. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα ε, εφόσον το πετύχει η Τραπεζική Ένωση. Τώρα για τη συγχώνευση των τραπεζών να διορθώσω λιγάκι γιατί αναφερθήκατε στη θέση μου αλλά εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θα ζητήσουμε κεφάλαια ε, σε περίπτωση συγχώνευσης. Αλλά υπάρχει μια αντίληψη στην αγορά ότι άπαξ και συγχωνεύονται δύο τράπεζες, αυτόματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ζητούσε αύξηση των κεφαλαικών απαιτήσεων. Πέρα δηλαδή από τις κεφαλικές απαιτήσει εφόσον ήταν χωριστά οι δύο αυτές τράπεζες πριν τη συγχώνευση. Αυτό όμως που λέω εγώ είναι ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά περίπτωση το σχέδιο συγχώνευσης και ποιο είναι το κεφαλαϊκό σχέδιο της νέας τράπεζες και να δούμε μεσοπρόθεσμα κατά πόσο υπάρχει διαδικασία που να επιτρέπει ε, την τήρηση των κεφαλικών απαιτήσεων. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κεφαλική θέση, γιατί συνήθως υπάρχει και μια αναδιάρθρωση όταν γίνεται συγχώνευση και μετά αρχίζει η κερδοφορία. Οπότε, εδώ, ο τραπεζικός τομέας έχει μεγάλη ικανότητα και κάποια συγκέντρωση πιθανόν να είναι καλή ιδέα. Όχι για να δημιουργήσουμε μεγάλους γίγαντες, αλλά μερικές φορές χρειάζεται η συγκέντρωση για να μην έχουμε πολύ μικρά μεγέθη. Μερικές φορές δεν είναι βιώσιμα αυτά τα πολύ μικρά μεγέθη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέντρο Μάρκες. Ευχαριστώ. Κύριε Ερία, για την ενημέρωση Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε δύο τμήματα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για το 2020 και πάλι είπατε να ε, καθαρίσουν οι ισολογισμοί των τραπεζών. Προφανώς το λαμβάνουν υπόψη αυτό οι τράπεζες για τις δραστηριότητες τους και αυτά που προβλέπουν για το 2020. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι τράπεζες έχουν περιέλθει σε μια ε, κατάσταση όπου έχουν περίπου 7% ε, απόδοση ε, και κέρδος συμμετοχές τους. Και αυτό φαίνεται και στον ισολογισμό. Μήπως να κοιτάξουμε περισσότερο τη την δομή των ισολογισμών και όχι την αποκατάσταση, το καθαρισμό τους. Για παράδειγμα, τα δάνεια σε ιδιώτες στα τελευταία στοιχεία έχουν αυξηθεί περισσότερο από ότι τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να αρχίσει ο υπόπτης να κοιτάει περισσότερο τη δομή την ίδια των ισολογισμών και τελικά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να δίνουμε τα σωστά κίνητρα για να υποστηρίζουν περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα οι τράπεζες και τις παραγωγικές επενδύσεις. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη, για την Τραπεζική Ένωση και την ολοκλήρωσή της. μας ανησυχεί λίγο ότι βρισκόμαστε πάλι σε ένα περιθώριο ε, καθημερινά κόκκινης γραμμής. Τελικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταφέρουμε τίποτα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι ότι έχουμε μειώσει πολύ τον κίνδυνο και χρειάζεται να ε, ολοκληρωθεί ο πυλώνας επιμερισμού κινδύνου, αλλά η τραπεζική ολοκλήρωση, η τραπεζική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να αντιμετωπίσει. Δεν είναι μόνο το Έντι. το Έντι είναι κρίσιμο. Ε, το θέμα των ασφαλών χαρτοφυλακίων ή της έκθεσης σε δημόσιο χρέος είναι σωστό, αλλά ε, είναι πάρα πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν μπορείτε αυτά να τα καταθέσετε ως προτάσεις ή σήμερα ή στο μέλλον να μας στείλετε τις σκέψεις σας. Ποια άλλα βήματα προτίθεστε να κάνετε για να ολοκληρωθεί πολύ περισσότερο ο τραπεζικός τομέας. Και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο έντις που είναι πολύ κρίσιμο, δεν αντιλέγω. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για το πρώτο που είπατε. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι. Εμείς είμαστε ε, προληπτική εποπτεία. Δηλαδή επικεντρωνόμαστε στον κίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασχολούμαστε μόνο ε, με ε, το καθαρισμό των ισολογισμών και των στοιχείων ενεργητικού που είναι κληρονομιά της κρίσης. Αν έρθει νέα ύφεση στις τράπεζες που ισχύει ακόμα στην Τραπεζική Ένωση. Έχουμε τράπεζες με 40% ή 30% κόκκινα δάνεια, μη εξυπηρετούμενα. Ε, θα, θα βρούμε πολύ σκούρα αν ξανάρθει η ύφεση. Κοιτάμε όμως τους κινδύνους και τα ρίσκα και σε άλλους τομείς. Αυτή τη στιγμή ε, που είναι χαμηλά τα επιτόκια, οι ε, τράπεζες διαφοροποιούν τα επιτόκια τους και ψάχνουν κερδοφορία από νέους ε, τομείς. Είπατε ότι αυξάνονται τα καταναλωτικά δάνεια, αλλά επειδή έχουν περισσότερο κίνδυνο καμιά φορά έχουν και μεγαλύτερη κερδοφορία. Δεν έχουμε δει αύξηση ε, στο δανεισμό μόχλευσης που μας απασχολεί πολύ επίσης. Δεν κοιτάμε μόνο τα χαρτοφυλάκια του παρελθόντος και την κληρονομιά που έχουν οι τράπεζες, αλλά και τους καινούριου κινδύνους που αναλαμβάνουν ε, και με αυτό μετράμε στον ε, τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται ε, οι τράπεζες. Είπατε πολύ διάφορα. Εμείς ως επόπτης δεν κάνουμε βιομηχανική πολιτική, μάλλον επενδυτική πολιτική. Δεν είναι δική μου δουλειά να δώσω κίνητρα σε μια τράπεζα να χρηματοδοτήσει τον α ή το β τομέα. Το θέμα είναι εμείς όταν παίρνουν αυτοί λάθος αποφάσεις να διαχειρίζονται σωστά τον κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση και ολοκλήρωση, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Πράγματι, έχουμε να αποθέσει πολλές ελπίδες στο έντις. Αν δεν έχουμε το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, αυτό χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να κατακαιρματίζεται ε, στις διάφορες χώρες η ρευστότητα και το κεφάλαιο. Γιατί αν πάει κάτι στραβά θα πρέπει το εθνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων να πληρώσει τα σπασμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα το έχουμε για κάποιο διάστημα ακόμα, γιατί το έντις δεν θα είναι έτοιμο από αύριο. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα ζητήματα και αρκετά που είναι και αντικείμενο νομοθετική συζήτηση. Είχαμε μακρές συζητήσεις ε, για ε, θέματα ρευστότητας και κεφαλαίων και με ποιο τρόπο διαχειρίζονται το ενεργητικό και το παθητικό τους οι τράπεζες ολοκληρωμένα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση, αλλά μιλάμε και ε, εδώ μιλικές εγγυήσεις. Ε, δηλαδή, εάν ε, μία θηγατρική ενός τραπεζικού ιδρύματος έχει πρόβλημα σε μία χώρα, η μητρική εταιρεία να το αναλάβει. Σε επίπεδο ομίλου δηλαδή να διαχειρίζεται. Και από πλευράς νομοθετικής προσπαθούμε να στηρίξουμε ε, αυτές τις λύσεις. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα μας βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντανούτα Χιμπνέ. Ευχαριστώ. Τρία ερωτήματα. Ε, πάνω σε πράγματα τα οποία έχετε ήδη αγγίξει, αλλά θέλω να τα διερευνήσουμε. Συμφωνώ καταρχάς μαζί σας ότι αν έχουμε ένα σχέδιο, ότι γίνεται μία ενιαία εναρμόνιση των εθνικών σχεδίων αφαιρεγγιότητας, χαθήκαμε. Ε, πρέπει να γίνει αυτό σε δόσεις, σε φάσεις και να δούμε τους τομείς όπου πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα ε, το να προτείνουμε μόνο ε, ένα σχέδιο για την ε, εκαθάριση είναι λάθος. Ε, ποιοι είναι αυτοί, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε δύο-τρεις τομείς για να ξεκινήσουμε με την εναρμόνιση, ε, για να την κάνουμε αυτή την εναρμόνιση βαθμιαία. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, σε διασυνοριακό επίπεδο, πώς θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεύτερο σημείο. Σχολιάσατε την Αμερική. Πώς αντιμετώπισαν την αντιμετώπιση της κρίσης στο τραπεζικό τομέα και πώς εκαθάρισαν τις τράπεζες. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ένα, είχαν μάλλον ένα κεντρικό εργαλείο και θα ε, θα, θα πρέπει να υπήρχε κάτι αντίστοιχο εδώ, ένα κεντρικό εργαλείο και στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας το αναπτύξετε λιγάκι περισσότερο αυτό το σημείο. Τρίτο σημείο, μιλήσατε για τις λιγότερο σημαντικές ε, οντότητες, τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, οι πιστοτικά ιδρύματα. Ε, ποιος είναι ο ρόλος σας ως επιποτική αρχή για αυτές τις τράπεζες. Κοιτάζετε τα πράγματα πιο συστημικά. Και πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το πλαίσιο της, ε, του εποπτικού μηχανισμού. Έχετε σκεφτεί καθόλου αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Για την αφαιρεγγιότητα. Θα απαντήσω στις δύο ερω... πρώτες ερωτήσεις μαζί. Καταρχάς, αν κοιτάξετε το τρέχον πλαίσιο για την ε, εξυγίανση των τραπεζών, την καθάριση των τραπεζών, έχετε κάποιες χώρες που έχουν διαδικασίες αφαιρεγγιότητας για τις τράπεζες, σαν να ήταν οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Δεν υπάρχει προστασία των καταθετών, δεν υπάρχουν διοικητικά εργαλεία, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε περιπτώσεις όπου στην ABNV, όπου ήταν μια τράπεζα που εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να χρεοκοπήσει γιατί είχε προβλήματα ρευστότητα. Μετά ε, Μία ανησυχία που είχαν εκφράσει οι Αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος ε, δεν μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία από το κράτος, ας πούμε, ε, για εκαθάριση. Έπρεπε να εθελοντικά η τράπεζα να κάνει τη δική της εκαθάριση. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουμε διοικητικά εργαλεία για την ε, καθάριση των τραπεζών, την νομοθεσία για την διαχείριση της αφαιρεγγιότητας τραπεζών ε, σε περίπτωση που υπάρχει τοπική διοικητική εκαθάριση, αυτή μπορεί να συνδυαστεί με κρατική βοήθεια. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα. Ε, είναι όμως πλατή. Θα πρέπει να το εναρμονίσουμε. Θα πρέπει να έχουμε ένα διοικητικό καθεστώς για την εκαθάριση τραπεζών, εκαθαρισμένο, ε, με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα έπρεπε οι αρχές να αναλάβουν ουσιαστικά, να ελέγχουν τις ε, προβληματικές τράπεζες. Μπορούν να το κάνουν λοιπόν αυτό. Οι καταθέτες ξέρουν ότι δεν πρόκειται να χάσουν ούτε ένα σέντ στην Αμερική από, το, από τα χρήματά τους, γιατί υπάρχει εγγύηση από, το, από τα κρατικά ταμεία των Αμερικανών. Ε, η τράπεζα αναδιαρθώνεται και ε, πουλούνται τα υπόλοιπα στοιχεία στις υπόλοιπες τράπεζες. Βγαίνει από τις αγορές, καθαρίζει τον ισολογισμό της κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και εμείς ένα τέτοιο εργαλείο. Υπάρχει και ενσωμάτωση, γιατί έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου ε, Εποπτικού Μηχανισμού και τότε δεν θα υπάρχει ε, διαφοροποίηση, ας πούμε, αναχώρα. Θα έχουμε μία πανευρωπαϊκή διαδικασία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το μέγεθός τους. Ε, κάνουμε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι, ότι παρότι η εποπτεία είναι στα χέρια των εθνικών αρμοδιών αρχών, ε, πρόσφατα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο το είπε αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμεί έχουμε μια συνολική ευθύνη για αυτέ τι τράπεζε. Δηλαδή, αλληλεπιδρούμε όλο και περισσότερο. Έχουμε ε, ε, διαιρέσει το μέγεθος ας πούμε, των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων ανάλογα με την προτεραιότητά τους, υψηλής προτεραιότητας, μεσαίας και χαμηλής κτλ. Και βεβαίως έχουμε αλληλεπίδραση ειδικά για τα πολύ κόκκινα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ας πούμε. Και συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές. Έχουμε μια συνολική προσέγγιση, συστημική προσέγγιση. Εξετάζουμε τη λειτουργία του μηχανισμού προστασίας των ε, ιδρυμάτων αυτών. Μερικές φορές εξετάζουμε το πώς λειτουργούν οι τράπεζες, τι ρόλο έχουν με βάση τα όσα διδαχθήκαμε την πρόσφατη κρίση και εναρμονίζουμε τα εποπτικά μας εργαλεία. Ε, εκδίδουμε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες μερικές φορές, αν χρειαστεί, προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν ορισμένους τομείς. Τη διαχείριση, ας πούμε, των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εκεί έχουμε πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα είμαστε, εξασφαλίζουμε ότι ε, εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές. Επίσης, ε, μερικές φορές ανακτούμε την εποπτεία. Αυτό έγινε φέτος ε, στην περίπτωση της ε, PNB, ε, μπάνκα της Λετωνίας. Αναλάβαμε την εποπτεία της τράπεζας, την αφαιρέσαμε από τις εθνικές αρχές. Και τώρα ε, θεωρούσαμε ότι είναι προβληματική, η τράπεζα βαίνει προς και της αφαιρούμε την άδεια σε αυτή τη φάση. Είναι ένα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από μερικές εβδομάδες ε, μιλήσατε για τη Βασιλεία Τρία στο, σε ένα τραπεζικό συνέδριο και απομακρυνθήκατε κάπως από την ιδέα ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα στις τράπεζες ε, για κεφαλοποίηση και ενεργητικό όπως επίσης και για το πράσινο ενεργητικό, γιατί είπατε ότι ο ρόλος σας είναι να είναι ασφαλέστερες οι τράπεζες και αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η έκθεσή τους σε κινδύνους. Σε άλλες συζητήσεις που είχαμε εδώ μαζί σας, είχατε αναγνωρίσει τους συστημικούς κινδύνους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όμως η συνέπεια των ε, φυσικών κινδύνων δεν νομίζω ότι πραγματικά αναγνωρίζονται. Είχαμε την ε, πρόεδρο Φοντερ Λάιεν χτε, η οποία ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μα μίλησε για τη Νέα Πράσινη Συμφωνία και για τι επιπτώσει που θα έχει αυτή σε όλου του τομεί τη κοινωνία. Οπότε, εμένα με απασχολεί το εξή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλε κεντρικέ τράπεζε ανά την Ευρώπη βρίσκονται στην αρχή ακόμα των δικών τους ευθυνών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτού στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εσείς επικεντρωνόσαστε ακόμα στη σταθερότητα και πώς θα αποφύγετε μια επόμενη κρίση σαν και αυτή που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι μηχανισμούς εσείς πιστεύετε ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να βοηθήσει το τραπεζικό τομέα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να μπει σε έναν πιο βιώσιμο δρόμο. Τι λέτε για την ε, έκθεση ε, σε κινδύνους για το κλίμα και τι θα κάνετε για να σωματώσετε τέτοια θέματα στην εντολή σας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι θα διευκρινίσω τα πράγματα. Γιατί πραγματικά δεν θα ήθελα να φύγετε και να έχετε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ασχολείται με μία από τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα είναι στην εντολή της ε, έκθεσης σύμφωνα με τη συνθήκη και θεωρούμε ότι είναι και δικιά μας εντολή να στηρίξουμε τους στόχους της Ένωσης. Οπότε οι περιβαλλοντικοί στόχοι και τα θέματα βιωσιμότητας βρίσκονται πάνω-πάνω ε, στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και τους δικούς μας. Το θέμα είναι ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής αλλά και στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των ε, αποκαλύψεων. Άπαξ και έχουμε την ε, ταξινόμηση του πράσινου ενεργητικού, τότε μπορεί το θέμα αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ τη βιωσιμότητα. Είδαμε πρόσφατα να κυκλοφορούν φήμες ότι οι τράπεζες σε κάποιες χώρες, ήταν πολύ φτωχές όσον αφορά ε, το πράσινο ενεργητικό του, τα διαπιστευτήριά του, τα πράσινα. Όλες αυτές οι τράπεζες λοιπόν εφόσον βγούνε και αποκαλύψουν στο δημόσιο τους πραγματικού τους στόχους, αυτό θα αποτελούσε ένα σημαντικό και δυνατό εργαλείο στη διάθεσή μας. Επιπλέον, με εργαζόμαστε πολύ για να δούμε τράπεζες θα διαχειριστούν τους κινδύνους τους που έχουν να κάνουν με κλιματικούς κινδύνους ή με πραγματικούς φυσικούς κινδύνους ε, σε σχέση με φυσικές καταστροφές ε, και λοιπά. Και αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ε, την οικονομία εφόσον υπάρξουν τέτοιοι κίνδυνοι. Και έπειτα είναι και το θέμα της μετάβασης. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ ε, όσον αφορά τις εποπτικές ε, προοπτικές, δηλαδή τι περιμένουμε εμείς από τις τράπεζες να κάνουν. Αν δέχεστε κάποιες εγγυήσει με δάνεια 25 ε, ετή, προφανώς και θα υπάρξει υποβάθμιση. Γιατί ας πούμε μπορεί να είναι ένα κτίριο το οποίο έχει αμίαντο. Οπότε τα, οι εγγύσει αυτές δεν πρέπει να κρίνονται μόνο με σημερινή αξία, αλλά να ληφθεί υπόψη και κατά πόσο τέτοιου είδους εγγύηση θα έχει αξία μετά από πολλά χρόνια. Ε, κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι θετικό όσον αφορά τη βιωσιμότητα είναι η χρήση των δοκιμών αντοχής. Αποτελεί κάθε τέτοια δοκιμή ένα σημαντικό ε, εργαλείο. Όταν ε, κάνουμε τις τακτικές τέτοιες δοκιμές, βάζουμε έναν ορίζοντα τριετή είναι πολύ δύσκολο όμως να καταλάβουμε τι θα έχει γίνει με τον κλιματικό κίνδυνο σε τρία χρόνια. Αν λοιπόν θέλετε να κρίνετε τα περιουσιακά στοιχεία, το ενεργητικό με σωστό τρόπο, τότε θα πρέπει να κάνετε και μια συγκεκριμένη άσκηση να λάβετε υπόψη σας μακροπρόθεσμα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν δουλεύει πάνω σε αυτό. Άρα ναι, βεβαίως. Τώρα η ερώτησή σας είναι ε, κατά πόσο οι κεφαλαιακές απαιτήσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ε, φορολογικό κίνητρο για να χρηματοδοτηθεί περισσότερο ένας κλάδος αντί για κάποιον άλλον. Τώρα, ανάλογα με τους κινδύνους θα δράσουμε. Πρέπει, αν μη τι άλλο, να αναλύσει κανείς σε βάθος ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι και μετά να αποφασίσει. Αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κανονικά, ο Σβέν Γκίγκολτ ε, έπαιρνε το λόγο, γιατί έχει γραφτεί και για δεύτερο. Ε, ωραία. Ε, εδώ λέει ότι θα παίρνατε εσείς το λόγο. Ε, το συζητήσαμε με το Σφέν και συγγνώμη που δεν σας ενημερώσαμε, ο κύριος Γιακελούνας. Αναφερθήκατε στις τράπεζες ε, FinTech που αυξάνεται αυτή η τεχνολογία χρηματοπιστωτική. Ε, τι γίνεται ε, με τις ε, ε, άδειες και κάποιους κινδύνους. Δίνετε κάποιες άδειες για τις τράπεζες FinTech, αλλά δεν έχετε εσείς την εποπτεία, την τακτική, την έχουν οι εθνικοί επόπτες. Και επειδή επικρεμάται τώρα και το Brexit, υπάρχει μια εποπτεία, εποπτεία και εμπορική δραστηριότητα ενδιαφέρον να ε, προσελκύσουμε κάποιες τράπεζες από τη Βρετανία. Εσείς το βλέπετε αυτό ως πρόβλημα ε, σε κάποια κράτη που θέλουν να προσεκίσουν τέτοιες τράπεζες fintech. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν εκδίδεται, εκδίδει την άδεια λειτουργίας ε, της τράπεζας αλλά την εποπτεία την έχει η Εθνική Εποπτική Αρχή. Ε, υπάρχει ηθικός κίνδυνος για μένα εδώ στην εποπτεία. Το θεωρείτε εσεί πρόβλημα ενδεχομένω ή όχι. Και αυτά τα δύο προβλήματα, και ο ηθικός κίνδυνος και ε, ο ανταγωνισμός ε, στην εποπτεία μπορεί να θέσουν προβλήματα στην ακαιρεότητα της αγοράς. Αυτό το παρακολουθείτε, το έχετε υπόψη σας, το θεωρείτε πρόβλημα, θεωρείτε ότι πρέπει να συζητηθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες επειδή στην Επιτροπή μας έχουμε στήσει και ομάδα εργασίας FinTech και το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να το παρακολουθεί τη CBA της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που καθοδηγεί τις τράπεζες για τις προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Απάντησε. Ευχαριστώ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θέτεται ένα πολύ ε, σημαντικό πρόβλημα. Όντως, βλέπουμε νέες τράπεζες να μπαίνουν στην αγορά που εκμεταλλεύονται νέες τεχνολογίες και όπως είπατε πολύ σωστά η διαδικασία του Brexit σημαίνει ότι πολλές τέτοιες εταιρείες FinTech ζητούν ε, να διοδοτηθούν ε, στην Τραπεζική Ένωση για να εξακολουθούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και μετά το Brexit. Το σημαντικότερο λοιπόν θέμα εδώ και το βασικότερο καθήκον για μας ήταν ε, η διαδικασία της αδειοδότησης. Αυτή είναι η δική μας αρμοδιότητα. Εμείς δίνουμε τις άδειες και πολύ σωστά είπατε ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο αδειοδοτήσεων για τις νέες ε, τράπεζες ε, τις ε, ψηφιακές fintech. Επίσης, δώσαμε μεγάλη έμφαση ε, στην εμπειρογνωμοσύνη που θέλουμε στη σύσταση των διοικητικών συμβουλίων τους, ε, ζητήματα όπως ε, εξωτερική ανάθεση του cloud, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και για τον Brexit. Λοιπόν, το πρώτο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο για την διοδότηση και νομίζω ότι αυτό το έχουμε στήσει. Όσο παραμένουν οι τράπεζες αυτές κάτω από το κατόφλι των σημαντικών των συστημικών τραπεζών, ε, η εποπτεία παραμένει στην Εθνική Εποπτική Αρχή. Την εκάστοτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται ή δεν το παρακολουθούμε. Ιδιαίτερα όπως σας είπα προηγουμένως, Έχουμε αρχίσει ένα τέτοιο διάλογο με αυτές τις εταιρείες, ε, κάναμε ένα ε, εργαστήριο και καλέσαμε αυτές τις ψηφιακές τράπεζες και τους επόπτες για να συζητήσουμε βασικά ζητήματα εποπτείας ακριβώς αυτού του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ε, κάναμε αυτό που λέγεται στα αγγλικά deep dive, δηλαδή έχουμε αναλύσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και θα τα εκδώσουμε όλα αυτά σε μια έκθεση που θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο. Γενικά, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το παρακολουθούμε είναι η κατάσταση μετά το Brexit. Να μην υπάρχει χώρος για εγκατάσταση κάποιων εταιριών που ε, θα αποφασίζουν εκείνες τι θα κάνουμε τους κανόνες και πώς θα τους εφαρμόζουν. Όχι, εφόσον οι τράπεζες εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα. Αν είναι εταιρείε παροχής χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών στο διαδίκτυο που δεν είναι τράπεζες και δεν έχουν άδεια τράπεζας, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και ενδεχομένω ε, εκεί αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA. Θα πρέπει όμως η νομοθεσία να είναι ουδέτερη τεχνολογικά και να ε, ισχύουν οι σωστές υποπτικές ε, ρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε διάει για λίγα λεπτά. Η κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Πολύ σοφή πολιτική. Να μην ε, θεωρήσουμε ότι οι πράσινες δραστηριότητες έχουν ε, επιβαρύνονται. Πρέπει όμως να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα μακροπρόθεσμα για το κλίμα και για την βιοπικιλότητα και, να... και για άλλους κινδύνους. Ε, ακούσαμε ότι η ΕΚΤ κάνει κάποια δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορείτε να σχολιάσετε τι σχέδια έχετε για να ενσωματώσετε ε, τον μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό κίνδυνο στην ανάλυση κινδύνου και στις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδεται προς τις τράπεζες, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες. Πότε, πώς εξασφαλίζουμε μια συνέπεια στις εκτιμήσεις μας. Όταν, όταν ας πούμε, να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικές δραστηριότητες. Την κυκλική οικονομία ή οποιασδήποτε άλλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τους ίδιους δείκτες. Ε, Βεβαίως υπάρχει και το μοντέλο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε πολλά μοντέλα. Πώς θα επιλέξουμε το σωστό. Ασχολούμαστε πολύ στο, με το δίκτυο ε, για, την, την, το πρασίνισμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ε, είμαι ένα από τα μέλη. Ε, είμαστε δραστηριοποιημένοι σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταλάβουμε τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και τους παράγοντες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Σε Μάλλον, να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ετοίμασε ένα οδικό χάρτη για κλιματικά θέματα. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και στηρίζουμε τη στρατηγική της, που έχει στοιχεία ε, αποκάλυψης, ε, ένα πλαίσιο για τις δοκιμές αντοχής και κατευθυντήριες γραμμές ε, προληπτικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να διαχειρίζονται σωστά τον κλιματικό κίνδυνο οι τράπεζες. Αυτό που κάναμε και που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι Κοιτάμε το δικό μας ε, το συγκεκριμένο προληπτικό στόχο. Έχουμε πάρει ένα δείγμα σημαντικών και λιγότερο σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συλλέγουμε στοιχεία για να δούμε κατά πόσο γνωρίζουν την, έκθεση, την έκθεσή τους ε, και την προσέγγιση τους τελικά στον κλιματικό κίνδυνο. Να δούμε πώς αντιμετωπίζουν τον ε, περιβαλλοντικό κίνδυνο. Έχουμε διάλογο, διάλογο με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές, με τις εθνικές αρχές και αναπτύσσουμε εποπτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τον κλιματικό κίνδυνο. Για να ενσωματώσουμε αυτό το στοιχείο, αυτό το κίνδυνο, ε, στο, στο εποπτικό πλαίσιο. Έχουμε ένα πλαίσιο με δύο πυλώνες, όπου κοιτάμε τη διακυβέρνηση, και βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο στο διοικητικό συμβούλιο τη τράπεζα που καταλαβαίνει από αυτά τα θέματα και πώ διαχειρίζονται αυτό τον κίνδυνο. Πώ επηρεάζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κεφαλαίου της τράπεζας. Αυτή είναι η εστίαση που έχουμε. Σε ό,τι αφορά την ε, γενική μας πολιτική, έχουμε ένα δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, όπου αλληλεπιδρούμε, συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για να λάβουμε υπόψη μας και να ενσωματώσουμε τον περιβαλλοντικό κίνδυνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους, που, όλους όσοι συμμετείχατε σήμερα σε αυτήν ε, την ε, συνάντηση και τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα περάσουμε στο σημείο 2 και 3 στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα όμως έχω να κάνω λοιπόν ανακοινώσεις όσον αφορά τις διαδικασίες ορισμών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, συμφώνησαν οι συντονιστές ε, για τους δύο υποψηφίους όσον αφορά τις θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου ε, να έχουν ακροάσεις με τους υποψηφίους και να ψηφίσουν στις, αυτό έγινε στις 3 Δεκεμβρίου. Έπειτα, όσον αφορά το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, συμφώνησαν οι συντονιστέ για τα επόμενα βήματα. Όσον αφορά την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή τη Συμβουλευτική Στατιστικών, ορίστηκε ο Βέρνερ Λάγκεν ω μέλο τη, θα οριστεί δηλαδή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω μέλο τη Επιτροπή αυτή, ο κ. Λάγκεν. Ομάδε εργασία τώρα. Μετά τη συζήτηση μεταξύ συντονιστών αποφασίστηκαν τα εξή. Τραπεζική Ένωση, Ομάδα Εργασίας. Έχουμε 22 μέλη. Ε, πρόεδρος της ΕΚΟΝΟ θα προεδρεύει. Ε, ανταγωνισμός. Έχουμε 12 μέλη και η Προεδρία πηγαίνει στο ΕΛΚ. Ε, χώρες πρόσβασης στο ευρώ, 12 μέλη και η Προεδρία πάει στους σοσιαλιστές. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 12 μέλη σε αυτήν την ομάδα εργασία και την Προεδρία την παίρνει το ΡΙΝΙΟΥ ομάδα εργασίας FinTech, 12 μέλη και την Προεδρία την αναλαμβάνουν οι πράσινοι. Ε, οι ομάδες πρέπει να στείλουν τα ονόματα που προτείνουν για την Προεδρία των ε, ομάδων εργασίας ε, στις οποίες θα προεδρεύουν. Μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου. Έπρεπε να είχε σταλεί τότε. Ε, ε, αναφορές τώρα. Άλφρετ Σάντ ορίστηκε για το δίκτυο των αναφορών. Οι ομάδες πρέπει να στείλουν ονόματα για αναπληρωματικά μέλη. Αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι την 21η Νοεμβρίου είχα πει, η συνέχεια για τις νέες αναφορές ε, που πήραμε στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών θεωρούνται εγκεκριμένες. Τώρα για το δίκτυο όσον αφορά το gender streaming. Μόνικα Σεμέντο από τη Renew ορίστηκε ως μόνιμο μέλος από πλευρά τη ΕΚΟΝΟ και η κύρα Πέτερ Χάνσεν αναπληρωματικό μέλος του δικτύου αυτού. Η οικονομική διακυβέρνηση τώρα. Πακέτο εξαμήνου. Εξετάζουμε ημερομηνίε τον Ιανουάριο για να έχουμε οικονομικό διάλογο με τους επιτρόπους όσον αφορά το πακέτο αυτό για το εξάμεινο. Επίσης συνάντηση εκόνο και προϋπολογισμοί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η πρόταση είναι για την 13η Ιανουαρίου στο Στρασβούργο και εγκρίθηκε αυτή η πρόταση. Έπειτα για την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα αποφασίστηκαν τα ε, για την οργάνωση που αναλαμβάνει ΕΚΟΝ για το πρώτο σκέλος προς ένα νέο διεθνές σύστημα φορολόγησης και θα έχουμε εκπρόσωπο από τον ΩΣΑ και ευρωβουλευτές και από τις χώρες ε, της Προεδρίας του 2020 προσκαλούνται. Δεύτερο σκέλος, από τη διαφάνεια στη βιωσιμότητα και στόχοι ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ θα έχουμε εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βουλευτές από την Προεδρία του 2020 ως ομιλητές. Και τελευταία ανακοίνωση για σχέδιο ψηφίσματος. Απασχόληση post-public, πώς θα αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, αφού κατέχει κάποιος κάποιο δημόσιο αξίωμα μετά τη πώς μπορεί να συνεχίσει τα διαδρομία του. Αυτά. Τώρα, για τριμερείς διαλόγους. Έχουμε έναν Econ NV για τις βιώσιμες επενδύσεις. Ε, και 5η Δεκεμβρίου έγιναν δύο τριμερεί διαλόγου και οι διαπραγματευτικέ ομάδε συμφωνούν επί τη αρχή όσον αφορά πολιτικά ζητήματα, κυρίω όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη χρήση των εκτελεστικών ε, και καταξουσιοδότηση πράξεων, τη δημιουργία επίσης ομάδας για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά και επίσης να συμπεραλάβουμε και δραστηριότητες μεταβατικές με την ε, ενημέρωση αποκάλυψη των υποχρώσεων. Επίσης τον αποκλεισμό των ορυκτών καυσίμων από τα κριτήρια ε, τεχνικού screening συνεχίζεται το έργο της ομάδας αξιωματούχων. Και τέλος, τριμερής διάλογος που έγινε ο τελευταίος, ήταν ο τέταρτος, χτες έγινε, στις 11 Δεκεμβρίου, όπου το Συμβούλιο είπε ότι ακόμα οι χώρες μέλη δεν έχουν ενημερώσει για τα διάφορα επίμαχα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα όρια και την περίοδο προβληματισμού. Υπήρχε προθεσμία μετά από το πρώτο μέρος του τριμερούς διαλόγου που θα ήταν τέσσερις το απόγευμα. Είχαμε έναν το πρωί και θα είχαμε άλλον έναν μετά τις 7 και είχαμε βάλει την προθεσμία λοιπόν στις 4 το απόγευμα για να έχουμε την αντίδραση του Συμβουλίου ε, και χρειάζεται πρόοδος ε, ο πρόεδρος όμως αποφάσισε να ακυρώσει το δεύτερο τμήμα του τριμερού διαλόγου γιατί δεν είχαν καταφέρει να λάβουν εντολή από τις χώρες μέλη. Οπότε η διαπραγματευτική ομάδα περιμένει τώρα από την Προεδρία του Συμβουλίου πριν ε, σχεδιάσει επόμενο τριμερή διάλογο. Περιμένουμε το Συμβούλιο λοιπόν. Τώρα. Χωρούμε στις ψηφοφορίες. θεσμικά όργανα και οργανισμοί στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσιο αξίωμα η υπηρεσία. Μια στιγμή να βρω ό,τι χρειάζομαι εδώ. Okay, let's first do a test. Να κάνουμε λοιπόν τώρα ένα δοκιμαστικό, μια δοκιμαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Everyone has voted. Ψηφίσατε όλοι. Δοκιμαστικά πάντα. Πέρασε. Okay. Good. So now we start. Ωραία. Αρχίζουμε την κανονική ψηφοφορία μας. Παράγραφος 1 του αρχικού κειμένου. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η δεύτερη παράγραφος. Η τροπολογία 9 και 10 που ταυτίζονται. Ε, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική τροπολογία α. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγραφός 4 του αρχικού κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβιβαστική τροπολογία C. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5 το αρχικό κείμενο ψηφί υπέρ, κατά, ε, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 6 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να το ελέγξουμε αυτό. Είναι η τροπολογία 25. Παρακαλώ. So, has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Μπορώ να κλείσω την ψηφοφορία, λέει. Υπάρχει ένας υπεράριθμος από την ομάδα Renew. Συγγνώμη, αλλά αυτό πρέπει να το λύσουμε κάπως. So, adopted. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 28. Όχι, διορθώνει η Πρόεδρος 26. Πέρασα την 26. Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα η τροπολογία 27. Υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 31 ψηφί υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 32 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 παράγραφος του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την αιτιολογική σκέψη, η αναφορά 1 έως 4 μαζί, υπέρ, κατά, citations, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πέντε με 11 υπέρ, αναφορές κατά αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αμπλοκ τώρα 12 με 17 αιτιολογικές αναφορές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις A ως D υπέρ κατά μαζί είναι όλες αυτές. Αποχές εγκρίνονται. Τώρα, συμβιβαστική F λατινικό. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 7 ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη I υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστικά παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Wow. Ομόφωνα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Just one minute. Ένα λεπτάκι. Okay, please, ladies and gentlemen, due to... Uh, Προέκυψε κάποιο ζήτημα με την πρόεδρο και μου ζητήθηκε να την αντικαταστήσω στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη, που είναι το σημείο 6, που είναι το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο με ιδιαίτερη χαρά στην εισηγήτρια, την Ινές Βάιντερε. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ας με προσέξουν λίγο συνάδελφοι, παρακαλώ, για να σας παρουσιάσω σύντομα την έκθεση αυτή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, οι επιχειρήσεις είναι προστιθέμενη αξία, αλλά έχουν και υποχρεώσεις να συλλέγουν το φόρο προστιθέμενης αξίας. Κάτι το οποίο βέβαια είναι μεγαλύτερο βάρος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από ότι είναι για τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις παρά τις εξαιρέσει που υπάρχουν για τι μικρές και μεσαίε επιχειρήσεις. Αυτό κυρίως ισχύει στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Στόχος της πρόταση αυτής λοιπόν τώρα είναι να τροποποιήσει τους κανόνες ε, ΦΠΑ ώστε να είναι πιο σύγχρονοι, ε, πιο απλοποιημένοι, να μειωθεί έτσι το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο στο εσωτερικό του, της κάθε χώρας όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι σημαντικό γιατί αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και πρέπει να απλοποιήσουμε όσο γίνεται την κατάσταση και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν περισσότερο και να δραστηριοποιηθούν και διασυνοριακά. Και άρα να δημιουργήσουν έτσι περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Αυτή η νομοθετική πρόταση λοιπόν ε, βρίσκεται στην διαδικασία ε, το, στην διαδικασία, λέγε, στο Συμβούλιο, ε, στη διαδικασία διαβούλευσης, ε, το Συμβούλιο ήρθε τον Νοέμβριο φέτος και αποφάσισε να ε, ξανασυζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον το κείμενο τελικά αλλάζει πολύ σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιανουαρίου που μας πέρασε. Για να επιτεθεί ο στόχος της πρότασης. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε διάφορα μέτρα τα οποία ε, διατηρούνται στην προσέγγιση του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, η μεταβατική περίοδος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς το συνδυσμένο ΦΠΑ ε, προεκτείνεται, παρατείνεται. Επίσης, η ιδέα του, της ενιαίας θηρίδας που βοηθάει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών ε, μελών ευθυγραμμίζεται και με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προηγούμενη έκθεση. Έτσι, συνεπώ, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, να διασφαλίσουμε ότι το βάρο για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει μειώνεται. Το Συμβούλιο, λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόσει όσο γίνεται πιο γρήγορα τους νέους κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν συμπεριληφθεί ε, στις ε, προδιαγραφές του Συμβουλίου, θα μπορούσε πολύ γρήγορα να προχωρήσει και να εξεταστεί και από το Συμβούλιο η έκθεση αυτή. Γι' αυτό και σας προτείνω την απλοποιημένη διαδικασία. Δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, οπότε πιστεύω ότι θα εγκριθεί στην πρώτη ολομέλεια του Ιανουαρίου η έκθεση αυτή στο Στρασβούργο. Και δεν ξέρω αν ε, θα μου δώσετε το λόγο ξανά μετά τη συζήτηση. Αλλιώς τώρα να ευχηθώ στους συναδέρφους καλά Χριστούγεννα, καλές διακοπές και κάθε επιτυχία για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Συγήτρια και σας ευχόμαστε και εμείς καλά Χριστούγεννα. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ε, σοσιαλδημοκράτες πρώτα, Αλφρέτ. Ευχαριστώ την ε, νέα εισηγήτρια για το φάκελο αυτό. Καλή, καλές ευχές και για τα Χριστούγεννα. Εξετάζουμε αυτή την πρόταση εκ νέου που θέλει να δώσει ευελιξία για το ΦΠΑ ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Σεπτέμβριο 2018 το Κοινοβούλιο με την έκθεσή του ενέκρινε το κείμενο. Πρότεινε οι μικρέ επιχειρήσει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την εξαίρεση στο ΦΠΑ για δύο ακόμα χρόνια, αντί για ένα χρόνο μόνο. Και όταν ξεπερνάει ο ετήσιος τζίρος το κατόφλι, να υπάρχει ένα, μια δικτυακή πύλη για να βοηθάει τις εταιρείες για αυτές. Ε, το Συμβούλιο με τις συντροποποίησεις του μειώνει το βάρος συμμόρφωσης, επομένως για να ενσωματωθεί γρήγορα ε, το κείμενο αυτό στην Εθνική Νομοθεσία θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο ε, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με το Συμβούλιο με το κείμενό του Νοεμβρίου του 2018. Πολύ ωραία. Καρολάιν, ε, Καρολίν, από το Ορνιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη θαυμάσια δουλειά. Το Συμβούλιο ε, ενέκρινε την ε, κοινή προσέγγιση τον περασμένο Νοέμβριο, γιατί περιμέναμε, περιμέναμε αρκετό καιρό την άποψή του. Και εγώ πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές ε, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα ειδικό σχήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους επιτρέπει αυτή τη στιγμή να υποφεληθούν από μία εξαίρεση. Η εξαίρεση στο κράτος μέλος όπου η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ε, δραστήρια. Όχι όμως εφόσον έχει διασυνοριακή δραστηριότητα. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε αυτό το φάκελο, ούτως ώστε και οι διασυνοριακές δραστηριότητες να υποφελούνται από την εξαίρεση ΦΠΑ. Γενικώ λοιπόν πώ και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησαν να μειώσουν το διοικητικό άχθο για τι επιχειρήσει και το κόστο συμμόρφωση για αυτέ τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. και πιστεύω ότι πραγματικά θα τι βοηθήσει αυτό το σχήμα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό το ειδικό σύστημα ελπίζω να είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, 100% υποστήριξη από πλευρά μου και συμφωνώ και με την απλουστευμένη διαδικασία. Και εγώ σα εύχομαι καλή τύχη και καλά Χριστούγεννα βεβαιω. Πάμε στους πράσινους. Ο ε, εκπρόσωπος, ε, εκπρόσωπος τους δεν είναι εδώ. Δεν θέλει κανένας να τον αντικαταστήσει. ID, κανένα εκπρόσωπο, ECR. Ο σχεδόν εισηγητής τους είναι εδώ. Ναι, είναι. Ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Τζουρτζίτσα. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Ε, μ' αρέσει εκείνη η προσέγγιση του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι η πρόταση θα βιώσει το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμφωνώ με, ε, με το αίτημα του Συμβουλίου να αντιδράσουμε το συντομότερο δυνατόν εμείς και να προχωρήσουμε την αποστευμένη διαδικασία. Ευχαριστώ. Γκουε. Υπάρχει εκπρόσωπο σκιώση ηγητή, δηλαδή, από την Γκουε. Όχι. Θα προχωρήσουμε την απλουστεμένη διαδικασία, χωρίς ε, τροποποιήσεις. Ε, ε, άρθρο 52.1. 28 Νοεμβρίου ήταν έτοιμο το σχέδιο αυτού του κειμένου. Και αν όλοι συμφωνείτε με αυτή τη ε, διαδικασία, γκρίνουμε με την απλή, απλουστευμένη διαδικασία, χωρίς τροπολογίες δηλαδή, το κείμενο αυτό. Ε, άρθρο 179, ε, αριθμός μελών 6 κάτω, ε, ή λιγότερα δηλαδή. Επομένως υιοθετείτε το κείμενο, εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, καλά Χριστούγεννα και στην εισηγήτρια λοιπόν. Η έκθεση λοιπόν θα πάει στην Ολομέλεια φυσικά από εδώ και πέρα. Now we can move to uh, item Πάμε στο 7. Δική μου έκθεση υποτίθεται. Αντικαθιστώ την πρόεδρο, τον πρόεδρο. Έχω διπλό λοιπόν ρόλο, διπλή ιδιότητα. που είναι προβληματικό για την πολιτική ανταγωνισμού. Προσοχή, προσοχή, γιατί η έκθεση αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. So λοιπόν. Θα μιλήσω για την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα μιλήσω γαλλικά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όλους και όλες αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίως τους κοιόδης εισηγητές με τους οποίους μπόρεσα να ξεκινήσω μια καλή συνεργασία ε, επί της εκθέσεως αυτής. Σίγουρα είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά είναι ζωτική σημασία για πολλούς λόγους, κυρίως για τρεις. Πρώτον έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια αντιπρόεδρο που είναι υπεύθυνη για τα ψηφιακά και τον ανταγωνισμό, ε, τη οποία γνωρίζουμε την αποφασιστικότητα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεύτερον, η πολιτική ανταγωνισμού τελικά έτσι όπως ε, έχει από την αρχή έπαιξε τον αρχικό της ρόλο, δηλαδή την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών με ελεύθερο ανταγωνισμό και όχι στρεβλωμένο μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επίσης βοήθησε και τον καταναλωτή να υποφεληθεί, αλλά υπάρχει συνειδητοποίηση γενικευμένη σήμερα και από πλευράς πολλών χωρών μελών και από τους πολίτες, αλλά εφ' και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι οι κανόνες ανταγωνισμού δεν προσαρμόζονται πλέον στον σημερινό κόσμο και δεν είναι και αρκετά αποτελεσματικοί για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Στη νέα μου έκθεση λοιπόν ήθελα να τονίσω τέσσερις άξονες που σίγουρα θα τροποποιηθούν και θα συμπληρωθούν στη συνέχεια, αλλά που κατά τη γνώμη μου αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες σε σχέση με τους οποίους πρέπει γρήγορα να δράσουμε. Πρώτος άξονας είναι ο ρόλος που έχει να παίξει η πολιτική ανταγωνισμού στην παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικός, να ενισχυθεί και να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που γνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε λόγω τη παγκοσμιοποίηση. Στην έκθεση αυτή ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει μια πιο συνολική προσέγγιση υπέρ της βιομηχανικής συνεργασίας για να επιτρέψει την ανάδυση Ευρωπαίων πρωτοκάθεδρων ανταγωνιστικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό και προτείνω αναθεώρηση του ορισμού της καλής αγοράς προκειμένου να λάβει υπόψη την παγκόσμια διάσταση και τον ε, ανταγωνισμό έτσι όπως πιστεύουμε ότι θα έχει στο μέλλον. Η κυρία Βεστάγκερ, η Επίτροπος, ε, συμφώνησε με αυτή την ιδέα και αποφάσισε να ξαναδεί την ανακοίνωση του 1997 σχετικά με αυτό τον όρο, ποια είναι δηλαδή η καλή αγορά, η αποτελεσματική αγορά. Έπειτα, για να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό και τις πρακτικές ε, τις σχετικές των επιχειρήσεων θα έπρεπε να ενισχύσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για τον έλεγχο των άμεσων επενδύσεων των απ' και ε, το θέμα της αμοιβαι... αμοιβαιότητας στις δημόσιες αγορές. Ε, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και σώροπη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Δεύτερον, τα ψηφιακά. Ε, δεν αποτελούν ένα ξεχωριστό τομέα, είναι χαρακτηριστικό της οικονομίας μας. Πρέπει τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Πρώτα απ' όλα, η τιμή δεν είναι η μόνη μεταβλητή για να κρίνουμε ε, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καταναλωτή, στην ευημερία του. Έχουμε και νέα στοιχεία τον 21ο αιώνα. Η διάσταση που συνδέεται με την ισχύ των αγορών και όλων των δεδομένων ε, είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει κάθε επιχείρηση συγκέντρωσης να ελεγχθεί προηγουμένως ανεξάρτητα από τα όρια και να υπάρξει αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για να αποφύγουμε τις λεγόμενες killer acquisitions. Και θα έπρεπε επίσης να εγκαθαρίσουμε και ε, μια διάταξη που να προβλέπει εξάντε ελέγχους των αγορών. Γι' αυτό και εκούρω τον κόδωνα του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συγκέντρωση δεδομένων προσωπικών και οικονομικών από κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κυριαρχούν στο τοπίο σήμερα και αυτό σε βάρος του ανταγωνισμού και του σεβασμού του ιδιωτικού βίου. Και γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Αρχή για την προστασία των καταναλωτών. Τονίζω επίσης και το θέμα των κυρώσεων. Οι κυρώσει είναι πρώτα απ' όλα πρόστιμα. Σοβαρά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι στοιχειώδες, αλλά δεν φτάνει. Γιατί μερικές φορές δεν τις νοιάζει τις επιχειρήσεις και τελικά την ύφη την πληρώνουν οι καταναλωτές. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερα ε, μέτρα ε, προστατευτικά, ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος των επιχειρήσεων. Και πρέπει επίσης να ε, διασφαλίσουμε ότι στοχεύουμε καλά το σύστημα και προηγουμένω να έχουμε συζητήσει με τις επιχειρήσεις που είναι θύματα μερικές φορές. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι αλλαγέ τις οποίες βλέπουμε σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε το κείμενο το οποίο εφαρμόζεται στις τομεκές πολιτικές στο μέλλον των αλλαγών που θα έχουμε στον ψηφιακό τομέα και την τεχνολογία. Και κυρίως να δώσουμε προτεραιότητα στους τομείς που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, την μετακίνησή του για παράδειγμα. Έπειτα, υπάρχουν οι κανόνε. Μίλησα πριν για τι κρατικές ενισχύσει. Αλλά και εδώ θα πρέπει οι κανόνες να λαμβάνουν υπόψη το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και οι σχετικές διατάξεις πρέπει να πλοπηθούν και να ε, μπορούν να λάβουν υπόψη και πολύ μικρά σχέδια και να υπάρχει επίσης και επένδυση στην, ε, στις τεχνολογίες ακόμα και την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Η έγκριση από την Airbus για τις ε, μπαταρίες είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσει πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται με την υλοποίηση και την εφαρμογή. Και τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει και πάλι το ρόλο του στην πολιτική ανταγωνισμού, η οποία όπως γνωρίζουμε, βρίσκεται κυρίω στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο που εκλέγεται απευθεία από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δυστυχώς πολύ συχνά ε, του ζητείται διαβούλευση. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει πιο ενισχυμένο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα του ανταγωνισμού, ενώ το Αμερικανικό Κογκρέσο μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και έρευνες για θέματα ανταγωνισμού. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε εμεί ε, ακριβώ τι ίδιε αρμοδιότητε με του Αμερικανού συναδέλφου μα, αλλά αν μη τι άλλο θα πρέπει να συμμετέχουμε πιο συχνά στα θέματα του ανταγωνισμού. Και τέλο, πρέπει να ανοίξουμε την πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και του βιομηχανικού στόχου, αλλά και του περιβαλλοντικού, γεωργικού, Έγινε να λάβουμε υπόψη μας το διεθνές εμπόριο, τους ε, κοινωνικούς μας ε, στόχους και οι εθνικοί ρυθμιστές και οι εθνικές ε, ομάδες καταναλωτών θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στο διάβημα αυτό. Πρέπει να πάψει να αποτελεί κλειστό σιλό όλη αυτή η υπόθεση του ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που με ακούσατε και χαίρομαι που μπορώ να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας και έτσι να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Και σε εσά εύχομαι καλά Χριστούγεννα, έτσι. So I now give the floor back to... Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο ε, και την Προεδρία στην αγαπημένη μας Πρόεδρο. Okay. Now I think we can uh, give... Ε, νομίζω ότι μπορώ να δώσω το λόγο τώρα στους Σκιώδης και αρχίζω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Λέω ε, ο κύριος Στέφαν Κιουκιμπέργκερ. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας αυτή που εξετάζουμε, το σχέδιο έκθεσης Ε, πολύ ωραία τα είπε η συγκήτρια. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κοινοβουλευτικής περίοδου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σωστό είναι αυτή τη στιγμή να δώσουμε νέες οθήσεις για την πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, το νιώθουμε όλοι μας. Ο κόσμος γυρίζει πιο γρήγορα, έχει επιταχυνθεί ε, ε, η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και στην οικονομία και στην πολιτική και θα πρέπει να αντιδράσουμε πολιτικά. Και νομίζω ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, ανακοινεί και σωστά πολλά θέματα και τα πολύ ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερα στο πρώτο τμήμα, όπου βλέπουμε ότι αλλάζει το παιχνίδι στον κόσμο μας, ιδιαίτερα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό δεν είναι χθεσινή εξέλιξη και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε ως Ευρωπαίοι σε αυτό. Σωστά λοιπόν ε, είναι αυτά που προτείνει η έκθεση. Η εσωτερική αγορά στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αφήνει μεγάλες εταιρείες πρωταθλητές να δημιουργούνται και να επιτρέπονται οι συγχωνεύσεις και οι συνεργασίες καλύτερα στο μέλλον για να μπορούν να δρουν και σε άλλες αγορές. Γιατί είναι παγκόσμιος ο ανταγωνισμός πια. Στη συνέχεια. Η πολιτική ανταγωνισμού μπαίνει και στα ψηφιακά ε, και τα αντιμετωπίζει καλά η έκθεση. Βεβαίως θα πρέπει ε, να ξανασυζητήσουμε τις λεπτομέρειες, ε, να δούμε πώς θα τις ρυθμίσουμε και επιφυλάσσομαι να το κάνω εξ ονόματος της ομάδας μου ή και προσωπικά. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο λεπτομερώς κάποια στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, ε, οι πάντες έχουν καταλάβει ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική ανταγωνισμού που να ε, μπορεί να δρά και πιο γρήγορα και πιο απλά και πιο αποτελεσματικά γιατί είμαστε πλέον στην ψηφιακή εποχή. Μ' αρέσουν και τα μέτρα που προτείνεται τα τομεακά. Προέρχομαι από μια περιοχή που εξαρτάται πάρα πολύ ακόμα από το λιγνίτη. Και αν θέλουμε, ας πούμε, στην περιοχή του Ρήνου, να ξεφύγουμε από το λιγνίτι και να πάμε σε άλλες μορφές ενέργειες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται κρατικέ ενισχύσει τα χρήματα που δίνει μια χώρα για να διαρθρωθεί μια περιοχή και να φύγει από τον άνθρακα. Αλλιώ πώ θα πετύχει η ενεργειακή μετάβαση. Επίσης χαίρομαι ε, και για το ρόλο που ζητάτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς θα το πετύχουμε αυτό να έχουμε διαφορετικό ρόλο. να μπορεί το Κοινοβούλιο να πλαισιώνει την ισχυρή κατά τα άλλα Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να γίνονται και οι συζητήσεις νυφάλια, αντικειμενικά, χωρίς συναισθηματικές φορτίσεις στο Κοινοβούλιο. Για θέσεις εργασίας και τα λοιπά, αλλά να κοιτάμε τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, θα βρούμε κάποιο τρόπο να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή και χαίρομαι για τη μελλοντική της επεξεργασία και τη συνέχεια που θα δώσουμε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα η Κάρμεν Καμπριέλα ε, Αβράμμα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αγαπητή εισηγήτρια, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω αυτή την έκθεση, το σχέδιο καλύτερα, είναι πολύ καλή βάση εργασίας. Είπατε ότι είναι έκθεση πρωτοβουλίας, είπε ο προλαλής σας. Ε, δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου, αλλά στέλνει πολύ χειρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ό,τι ψηφίσουμε ε, τον Απρίλιο ή τον Μάιο θα είναι ισχυρό μήνυμα και ισχυρό και δεν μπορεί να το αγνοήσει η Αντιπρόεδρος Βεστάγκερ. Είναι ε, νέα η εποχή μας, ψηφιακή, με πάρα πολλές προκλήσεις. Αρχίζουμε από την Ευρωπαϊκή Νέα Πράσινη Συμφωνία. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις αναθεωρούνται και ελαστικοποιούνται. Για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη που θέλουν να δώσουν ενισχύσει για πράσινα βιώσιμα έργα ε, που θέλουν να φτάνουν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Ξέρω ότι πολλά μέλη της δικής μου πολιτικής ομάδας ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παρακολουθούμε και τις ενδεχόμενες ανητικές παρενέργειες. Κάποιες μεγάλες εταιρείε μπορούν να πρασινίσουν αλλά και μετά μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις ε, κρατικές ενισχύσεις για αλότριους σκοπούς στην περίπτωση της Αλιτάλια, ας πούμε, είναι θεμητά και εύλογα τα ερωτήματα σχετικά με την ε, ε, εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. 900 εκατομμύρια τους δώσανε. Ξεκίνησε μια υπόθεση πέρυσι στο δικαστή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα βλέπουμε ότι δώσαν και άλλα 400 εκατομμύρια χωρίς καν αυτό να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρα πολύ κακό προηγούμενο για άλλες εταιρείες που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ε, και θα μπουν στον πειρασμό να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαφανθεί πολύ σύντομα γι' αυτό, γιατί θα υπάρξει χιονοστιβάδα που θα μεγαλώνει συνεχώς. Για τις περιπτώσεις κατά των συγχωνεύσεων και των τραστ, ε, το θέμα της ταχύτητας είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε την υπόθεση Google Shopping που έχει αρχίσει, ανοίξει πριν από 10 χρόνια. Ψηφιοποίηση σημαίνει ότι οι αγορές κινούνται ραγδαία θα πρέπει και εμείς να επιταχύνουμε και να βελτιώσουμε ε, τις ε, περιπτώσεις καταπολέμησης διαφόρων ε, τράστιν. Τα δεδομένα είναι το σημερινό χρυσάφι. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες υπηρεσίες που προσφέρουν διάφορες πλατφόρμες. Πληρώνουμε ένα πάρα πολύ ψηλό τίμημα που είναι τα ίδια μας τα προσωπικά δεδομένα έχουν ξεσπάσει κάποια σκάνδαλα και τώρα έχει καταλάβει περίπου ο κόσμος τι συμβαίνει, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγκόμουνου. Θέλω να επιμείνω σε αυτό. Να το κοιτάξουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα προστασίας ιδιωτική ζωής, δεν είναι μόνο θεμητό, αλλά είναι και ανάγκη να ε, αναθεωρήσουμε τους κανόνες και τα εργαλεία ε, του ανταγωνισμού για τα δεδομένα. Είπε η κυρία Βεστάγκη ότι θα αναθεωρήσει τον όρο αγορά. Δεν είναι μόνο γεωγραφικός όρος. Είναι νέες οι προκλήσεις. Είναι δύσκολο από τους καταναλωτές να περάσουν από ένα οικοσύστημα σε ένα άλλο. Ε, έχουμε μια ψευδέστηση ότι επιλέγουμε αλλά καμία σχέση. Μπορούν κάποια οικοσυστήματα να εγκλωβίσουν κάποιους καταναλωτές. Ε, υπολογίζουν το κόστος οι μεγάλες εταιρείες τα, ε, και τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές δεν θέλουν να τα χάσουν οι μεγάλες εταιρείες. Ε, θα πρέπει να δούμε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τις αλλαγές ε, και της δομής και της συμπεριφορά έχουμε τις ευκαιρίες, έχουμε τροπολογίες που ζητούν περισσότερους εκπυρογνώμονες στην τεχνητή νοημοσύνη και μηχανικούς ε, υπολογιστών για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτά τα συστήματα. Σε άλλους κλάδους ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το τραπεζικό σύστημα στη Ρουμανία, όπου οι καταναλωτές βλέπουν ψηλά επιτόκια και αδιαφάνεια ε, για τις χορηγήσεις όταν ζητούν ε, δάνειο. Υπάρχουν απάτες ε, στην πώληση ε, τέτοιων δανείων και ε, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δύο φορές έχει αναφέρει αυτό το πρόβλημα της Ρουμανίας το 2018 που έχει τη μεγαλύτερη απόκληση στα επιτόκια δανεισμού. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει την ισχύ που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και επίσης ε, ε, για το πώς ε, διαμορφώνουν τις τιμές των παραγωγών. Οι παραγωγοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν παράπονα. Ακόμα και για τον τρόπο και τη θέση στο ράφι που βάζουν τα προϊόντα τους στο σούπερ μάρκετ. Επίσης για τις χώρες Μερκοσούρ θα έρθουν να μας κατακλείσουν διάφορα προϊόντα χαμηλότερου κόστους που δεν ε, πρέπει να σέβονται τα ίδια πρότυπα και προδιαγραφές και μπορεί αυτό να πυροδοτήσει αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Εγώ ε, ε, ζητώ ένα πιο διαρθρωμένο και τακτικό διάλογο με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και την κυρία Βεστάγκερ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμεσα εκπροσωπεί ακριβώς τους 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές και θα πρέπει να θεωρείται προνομιούχος συνομιλητής, τουλάχιστον περισσότερο από ό,τι σήμερα από τη ανταγωνισμού. Ευχαριστώ και προσβλέπω να συνεχίσω την επικοδομητική συνεργασία με όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικά, στο σχέδιο έκθεσης, για το οποίο ευχαριστούμε την εισηγήτρια, υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα θέματα που μας αρέσουν και μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με πνεύμα συμβιβασμού. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η εισαγωγή είναι πολύ γενικόλογη. Γιατί αν η αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού είναι βάρος στους ανταγωνιστές, ας πούμε, που ανταγωνίζονται σε παγκόσμια αγορά, αυτό το, το εκφράζει ως αρχή. Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο είναι σωστό μόνο εάν έχεις ε, τομεί ανταγωνισμού θα είσαι ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά. Δεν είναι βάρος η πολιτική ανταγωνισμού για όλες τις ανταγωνιστικές εταιρείε. Και σε μελλοντικού τομεί όπω η ψηφιοποίηση και το πρασίνισμα τη οικονομία ήταν ακόμα πιο αληθέ αυτό. Επομένω, δεν πρέπει να δείξουμε αυτή την αφέλεια Φυσικά πρέπει να υπάρξουν όρια, συμφωνώ με αυτό, αλλά μια γενική έκκληση να έχουμε μια ισορροπημένη εφαρμογή ε, στο σημείο 5 ε, των, κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι μια πολύ γενικόλογη αμφισβήτηση όλων όσων έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Έχουμε μια κοινή αγορά με 500 εκατομμύρια πελάτες, καταναλωτές μας δίνει ευκαιρίες αυτό. Να έχουμε ανταγωνισμό. Αν είναι λειτουργική η ενιαία αγορά, προς όφελος ακριβώς των καταναλωτών, προς όφελος των οντοτήτων και φορέων και εταιριών που μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια, στην παγκόσμια αγορά. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιοι τομείς που πρέπει να μας απασχολήσουν πιο συγκεκριμένα και πιο ειδικά. Ε, περιπτώσεις συγχωνεύσεων και περιπτώσεις ας πούμε, κρατικών ενισχύσεων που όντως μπορούν να στρεβλώσουν το διεθνή ανταγωνισμό. Αλλά θα πρέπει να περιοριστούν ε, και θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε αυτά με λεκτικό, ε, μονοσήμαντο τρόπο. Δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιε γενικόλογε διατυπώσει που αμφισβητούν ακόμη και διατάξει συνθήκη. Ό,τι αφορά το πρασίνισμα τη πολιτική ανταγωνισμού, έχουμε κάποια φρασιολογία που έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτή. Δυστυχώ η Κομισιόν δεν ήταν πολύ θετική σε όλα τα προβλήματα που είχε το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να ξανατονίσουμε κάποια από τα θέματα όπου η Κομισιόν δεν απάντησε θετικά στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Είμαστε θετικοί στην ιδέα σας για ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της αγοράς εκ των προτέρων, επίση ένα φορέα προστασίας των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο ισχυρές δραστηριότητες για τις πλατφόρμες στο ψηφιακό τομέα. Επίσης να υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο κοινοβούλιο τόνισε τα προβλήματα που είχαμε και που έχουμε ήδη και τώρα στην αγορά του τουρισμού το 15% των ξενοδοχείων σε, στην Ήπεθρο ε, υποκαθιστούνται από τους παρόχους ε, και διαχειριστές ε, πλατφορμών. Και αυτό στερεί ε, έσοδα από τις περιοχές της Ήπεθρο αλλά και, τις, και στις πόλεις όπου πηγαίνουν σε διάφορες .com. Έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο στην αγορά που τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια ε, δεν μπορούν να αποφύγουν αυτές οι πλατφόρμες. Η Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτεί πως πρέπει να βάλει ανώτατα όρια στις τιμές. Γιατί πραγματικά αυτές οι πλατφόρμες ε, εκμεταλλεύονται ε, τους κανόνες στον τομέα τον ψηφιακό. Τους δίνει πλεονέκτημα βεβαίως στην αγορά, αλλά θα πρέπει να τις οδηγήσει και σε καθαρή κλοπή. Επίσης, στην ενέργεια και στην πολιτική του ανταγωνισμού που τη αναφέρετε, θα πρέπει να είστε πιο συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να πείτε, ε, στα πλαίσια της ε, πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να θεωρήσουμε του κανόνε των κρατικών ισχύσεων, ούτω ώστε η ενέργεια που παράγεται από του καταναλωτέ εξαιρείται ε, από του δημόσιου διαγωνισμού. Επίση, η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με τι άλλε μορφέ ενέργεια. Τέλο, είναι ε, για αναθεώρηση της γενικής εξαίρεση σε ό,τι αφορά την αυτόματη εξαίρεση των περιφερειακών αεροδρομίων που οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των ε, ενισχύσεων για μη λειτουργικά αεροδρόμια, προβληματικά ας πούμε περιφερειακά αεροδρόμια. Ο Ντέρ Κέπινγκ. Δεν σας είχα δει, συγγνώμη. Ε, ναι, κάθομαι τόσο μακριά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεση που είναι καλή βάση για διαπραγμάτευση. Θα περιοριστώ σε λίγα σχόλια σε τομεί όπου θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε βελτιώσει. Πρώτον, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σεβαστούμε την ανεξαρτησία τη Γενική Διεθνή Ανταγωνισμού ε, για την εκτέλεση και την εφαρμογή της πολιτική ανταγωνισμού. Το Κοινοβούλιο πρέπει να πει την άποψή του για τη γενική πολιτική ανταγωνισμού, αλλά δεν θα πρέπει να προδικάζει με μονομένες και συγκεκριμένε περιπτώσεις. Θα προτιμούσα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη στυλίτευση συγκεκριμένων εταιριών στα πλαίσια της έκθεσης. Διαφωνώ επίσης με την έκκληση για να έχει ερευνητικές εξουσίες το Κοινοβούλιο, όπως ας πούμε έχει το Κογκρέσο στις ΗΠΑ που έχει τελείως διαφορετικές αρμοδιότητες και άλλο, άλλη δομή. Επίσης, μας αρέσει η διατύπωση για την φορολογία στο σχέδιο έκθεσης. Η φορολογία μπορεί να προκαλέσει θέματα και προβλήματα ανταγωνισμού. Με την ετήσια έκθεση ανταγωνισμού, η ετήσια αυτή έκθεση δεν θα πρέπει να γίνει έκθεση για το, τη φορολογία. Και ευχαριστούμε την εισηγήτρια που δεν μπαίνει στα χωράφια του, της φορολογίας και περιορίζεται στο πεδίο του ανταγωνισμού. Ε, όμως σε άλλες παραγράφους δεν έχουμε σωστή εστίαση. Ε, οι, παρά... οι παράμετροι της πολιτικής ανταγωνισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν ισοτιμία για τις επιχειρήσεις μεγάλες ή μικρές. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε υπερβολικά τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού με άλλους στόχους πολιτικής, παραδείγματο χάρη οικολογικούς ή κοινωνικούς στόχους. Είμαστε σκεπτικιστές ό,τι αφορά την έκκληση για τη δημιουργία νέων οργανισμών ή νέων φορέων. Θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα και πιο πιστικά επιχειρήματα πριν δημιουργήσουμε ένα μια Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Καταναλωτών. Κλείνοντα. Η εισηγήτρια γνωρίζει τα θέματα γιατί ήταν ε, δικηγόρος ε, για θέματα ανταγωνισμού. Τη συγχαίρω, αλλά θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση είναι καλή βάση διαπραγμάτευσης και ο κύριος Βίτο, ο σκιώδης ε, του ECR, θα υποβάλει επικοδομητικές τροπολογίες, ούτως ώστε να φτάσουμε σε συμβιβασμού που θα τη στηρίξει μια πλατιά πλειοψηφία. Έχω και μια τελική ερώτηση. Είναι θέμα διαδικαστικό. Σήμερα έχουμε 12 Δεκεμβρίου. Ε, στον τύπο διάβασα ότι η συγγύτρια παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης στην Επίτροπο Βεστάγκερ στις 6 Νοεμβρίου, πριν, 26 Νοεμβρίου, πριν δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες πριν μας την παρουσιάσει εδώ ίσως δεν γνωρίζω αρκετά τις πρακτικές. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν διαφορετικούς ρόλους όμως. Λοιπόν, το ερώτημα μου είναι, είναι σωστό η έκθεση να παρουσιάζεται πρώτα στην Επίτροπο πριν παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Θέλω να με φωτίσετε και να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις, αγαπητή συγγήτρια, για τα διαδικαστικά αυτά θέματα. Ε, Ευχαριστούμε. Ε, Μανώνο Μπρι. Καλημέρα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πρώτη αυτή εκδοχή. Υπόθηκε ότι είναι ιδίας πρωτοβουλίας, δεν είναι νομοθετική έκθεση αυτή, αλλά είναι σημαντικό παρόλα αυτά να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού που είναι τόσο βασική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπατε κι εσείς στην παρέμβασή σας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό διακύδευμα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και παρά το περιορισμένο πεδίο της έκθεσης αυτής, θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια σημεία και εγώ γι' αυτό θα τα συνοψίσω σε τρία. Πρώτον, οι κρατικέ ενισχύσει, που είναι και επικαιρότητα, γιατί αποτελεί μέρο τη Πράσινη Συμφωνία που μα παρουσίασε η Ursula von der Leyen χτε η προηγούμενη επιτροπή είχε ξεκινήσει μία αξιολόγηση για, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και είναι σημαντικό με τις κρατικές αυτές ενισχύσεις η αξιολόγηση να αναλύσει τι επιπτώσει που έχουν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντο τη δημιουργία μακροχρόνιων θέσεων απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων. Επίση θα έπρεπε να αξιολογηθούν και να θεωρηθούν και οι κανόνε που έχουν να κάνουν με το κοινό συμφέρον και να βελτιωθούν οι μεταφορέ, οι κοινωνικέ κατοικίε κλπ. Θα έπρεπε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι σημερινοί κανόνε είναι συμβατοί με του στόχου αυτού και να διευρύνουμε τον ορισμό των κρατικών ενισχύσεων. Δεύτερον, το θέμα της φορολογίας. Μετά από τον προλαλήσαντα, η πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού έχει να κάνει με τη φορολογία. Γιατί τα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρονται, χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες, τα εκμεταλλεύονται θα το έλεγα πιο σωστά, οι μεγάλες πολυεθνικές και οδηγούνται σε το ανταγωνισμό σε βάρος των ε, μικρότερων επιχειρήσεων. Το θέμα το φορολογικό φύγεται στην έκθεση, αλλά πολύ λιγότερο από ό,τι σε προηγούμενες εκθέσεις των προηγούμενων ετών και δεν Υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το θέμα του αθέμετου ανταγωνισμού εξαιτία της φορολογίας. Δεν αναφέρεται ε, ως αθέμετος ανταγωνισμός η φορολόγηση αυτή σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκθέσεις. Στο θέμα της ε, διαφάνειας το Συμβούλιο επίσης δεν κατάφερε να βρει λύση. Διχάζεται όσον αφορά την φορολογία. Υπάρχει έκθεση του ΩΣΑ, ε, υπάρχει και το σχέδιο τάξη της ΕΚΤ και οι πρώτοι που θίγονται είναι οι μικρές επιχειρήσεις βέβαια που δεν έχουν θηγατρικές σε οικονομικούς παραδείσους όπως μπορεί να είναι η Ιρλανδία ή αλλού. Συνεπώς, θα έπρεπε να τα υπογραμμίζει όλα αυτά η έκθεση και να κάνουμε όπως και με τις προηγούμενες εκθέσεις, δηλαδή να υπάρξει αναρμόνιση από πάνω στον φόρο των επιχειρήσεων, να βρεθεί μια λύση για το θέμα της φορολογίας, να προχωρήσει το θέμα του άξης επίσης ώστε να λυθεί και να προωθηθεί περισσότερο και να προχωρήσουμε και με τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσεων για να τηρηθούν τα κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες μέλη για να υπάρχει συνοχή και τα φορολογικά πλεονεκτήματα να μην προσφέρονται ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, κάτι άλλο που δοθεί η έκθεση είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός εξαιτία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τρίτε χώρε. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει κοινωνική εναρμόνιση στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν διαφορετικέ νομοθεσίε οι διάφορε επιχειρήσει, όπω γίνεται και στο φορολογικό. Και θα έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση για τον ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό να προχωρήσει και να εφαρμοστεί παντού στην Ευρώπη. Και παρόλο που τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουμε ε, για προστασία από τον αθέμητο ανταγωνισμό δεν θα έπρεπε τα περιβαλλοντικά μέτρα να ε, δρούν τιμωρητικά σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Από τη μια εμείς δυσκολεύουμε την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά επιχειρήσεων που βρίσκονται σε χώρες που δεν τηρούν ε, του, τις ρυθμίσεις για τα εργασιακά. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε ελεύθερες συναλλαγές με την Ιαπωνία για παράδειγμα που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αξιολογεί τις επιπτώσεις κάθε φορά που αλλάζουν οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί κανόνες σε μια χώρα και το είπε και η συνάδελφο από του σοσιαλιστέ ε, νωρίτερα, οι ελεύθερε συναλλαγέ με τη Μερκοσούρ είναι ένα άλλο παράδειγμα, όπου η Βραζιλία επιτρέπει φυτοφάρμακα ε, σε προϊόντα τη που εισάγει η Ευρώπη. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε αυτού του νέου κανόνε και να προταθεί μια αναθεώρηση που να είναι συμβατή και με την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία που μα παρουσιάστηκε χτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα, ε, επειδή έχουμε κάτι δύο αιτήματα, να δώσουμε το λόγο σε αυτούς τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο Αν δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, ε, και επειδή περιμένω πολλή ώρα, θέλω να, να μιλήσω. Έχω πολλά θέματα να πω. Πρώτον, χαίρομαι που η συγγήτριά μας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας προσπάθησε να μην πέσει στην παγίδα να χειραγωγήσει την έκθεση αυτή για ίδιους πολιτικούς σκοπούς, σκοπιμότητες. Αυτό πάντα γίνεται με την πολιτική ανταγωνισμού και αν θέλει το κοινοβούλιο να το παίρνουν πιο σοβαρά, να μην το κάνουμε όπως το κάνουν οι πράσινοι που θέλουν πιο πράσινισμα και κάποια άλλη άλλα πράγματα. Η πολιτική ανταγωνισμού υπάρχει για να εξασφαλίζει ίσους κανόνους παιχνιδιού στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και αυτό είναι αρκετά σκληρό για τις εταιρείε. Όλα τα υπόλοιπα λύνονται αλλού. Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, αλλά όπως είπε κάποιος άλλος συνάδελφος, αυτό θα γίνει μόνο αν τηρούμε τους κανόνες. Και χαίρομαι που αναφέρθηκε στις μπαταρίες ε, η συγγετρία που εγκρίθηκε αυτή η κρατική ενίσχυση τη Δευτέρα, τούτη την εβδομάδα. Στο Φέσενχάιμ θα κλείσει το πυρηνικό εργοστάσιο και γι' αυτό εγκρίθηκε η συγκεκριμένη ενίσχυση. Το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε η Επίτροπος ότι θα αλλάξει ε, τον ορισμό της αγοράς Ιδιαίτερα για τι συγχωνεύσει είναι αυτό σημαντικό. Ελπίζω να έρθει η Επίτροπος να μας εξηγήσει τι αλλαγέ θα κάνει έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε καλύτερα και σφαιρικότερα να αξιολογούμε τι συγχωνεύσει που θα γίνονται. Ένα παράδειγμα που βλέπω ε, με πολύ κριτικό μάτι ήταν ε, η ε, συγχώνευση ε, της MXP με την άλλη εταιρεία που ήθελε. Πληρούσαν όλες τις διατάξεις για τις συγχωνεύσεις και τον ανταγωνισμό, αλλά δεν έγινε δυνατή αυτή η συγχώνευση, διότι οι κινέζικες αρχές θεώρησαν ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε ε, άλλες ε, χώρες να αποφανθούν για δικές μας συγχωνεύσεις. Θέλω να επανέλθω στα τραπεζικά που ανέφερε η Κάρμεν Αβραμ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Παντού ένα άρθρο των Financial Times έλεγε πριν από 15 μέρες ότι αποφάσισε η Google να συνεργαστεί με τη Citibank. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Έχουμε πάρα πολλές τράπεζες. Δεν επιτρέπεται τώρα ένα ε, ε, μονοπόλιο να μας έρθει και να αποφασίζει για τους πολίτες. Και τελειώνω, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον ε, Dirk Epping και χαίρομαι που τον βλέπω εδώ σήμερα. Δεν θα πρέπει να κατονομάζονται εταιρείε ρητά στην έκθεση, να το περιγράφετε με τρόπο που να είναι σαφής, αλλά για να μην υπάρξουν παρερμηνίες ή καταχρήσεις του κειμένου, μην λέτε εταιρείε ονόματα. Ευχαριστώ. Ο Πολ Τάνκ, δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο ΚΑΤΣΙΑΙ, να γίνει ευρύτερη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και το εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως και ο Ανδρέας Φαπ. Σε ευχαριστώ, Στεφανή. Πολύ ενδιαφέρουσα ε, η συζήτηση και η έκθεση. Γενικά, η πολιτική ανταγωνισμού είναι στην καρδιά, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ε, εσωτερικής αγοράς. Υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει πάντα να βλέπουμε ποιος είναι ο ορισμό της αγοράς όταν είναι παγκοσμιοποιημένη οικονομία φυσικά. Αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις συγκεντρώσεις ε, της ισχύω στην αγορά. Αυτό είναι η ουσία βασικά, να υπάρχουν οι κανόνες παιχνιδιού. Μια γενική παρατήρηση έχω. Αναφέρθηκε ο Σφεν Γκίγκολτ στην παράγραφο 5, αλλά υπάρχει και παράγραφος 6 για την ε, βιομηχανική συνεργασία. Ε, τι θέλουμε, περισσότερη συγκέντρωση ή να αποφύγουμε τη συγκέντρωση και την ε, υπερισχύ στις αγορές. Θα πρέπει να είναι αυστηρή η πολιτική ανταγωνισμού, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους και αυτό να παραμείνει ως γενικό σχόλιο. Δεύτερο, για τη φορολόγηση ένα πιο ειδικό. Επαναλαμβάνει ότι καμιά φορά χρησιμοποιείται η φορολογία ως έμεση κρατική ενίσχυση. Χρησιμοποιείται καμιά φορά. Πολύ μαλακά τα λέτε. Υποτιμάτε την κλίμακα. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από τις Ολλανδικές πολυεθνικές που δεν πληρώνουν φόρο και δεν παίρνουν και κρατικές ενισχύσεις καν. Όχι όλες, εν πάση Φυσικά δεν υπάρχουν κανόνες ε, ε, καλού ανταγωνισμού και υγιούς μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών ε, επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει και περισσότερο λόγο και ρόλο. Ένα τελευταίο. Αυτό το ταμπού που δεν αναφέρει κανείς. Ξέρουμε ότι στις ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχει συγκέντρωση. Μπορεί να μην με αφήνετε να μιλήσω για την Google ή το Facebook. Γιατί είναι ταμπού, δεν το, το βλέπουν όλοι και δεν το αναφέρει κανείς. Ε, στην ακρόση της κυρίας Βεστάγκερ τη ρώτησα ξανά. Ε, τι θα κάνετε, θα, θα, θα προσφύγετε εναντίον τους. Ε, λέει είναι μία από τα, τις δυνατότητες που έχω. Γιατί και ποιες άλλες έχετε. Είναι πολύ μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς και εκεί πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να αναπτύξει κανείς ευρωπαϊκή εναλλακτική πρόταση. Και αυτό έχει να κάνει και με τις εξωτερικότητες του δικτύου. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα πρέπει να σκεφτεί ιδέες που μπορεί να είναι ε, η φορητότητα των δεδομένων από τη μια πλατφόρμα στην άλλη ή να υπάρξει απαγόρευση κάποιου είδους ε, ε, προσωπικών αγγελιών κτλ. Αλλά είναι μεγάλο ταμπού και δεν το συζητάει κανείς. Γιατί, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, μια που έχουμε εδώ τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, την κυρία Βεραρέχο, που ασκεί καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας. Ε, θα, με ενδιαφέρει να την ακούσουμε. Παρακαλώ. Α, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντινάκλη. Έχω σχόλια και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την πρόσκληση. Και πραγματικά είμαι ειλικρινής όταν σας λέω ότι με εκπλήσω ο βαθμός στον οποίο κατανοείτε την πολιτική μας. Γιατί αρκεί να ακούσει κάποιος αυτά που λέτε εδώ στη συζήτηση αυτή της έκθεσης για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Μπορεί να είναι περιττό, αλλά θα σας το πω παρόλα αυτά, ότι η Αντιπρόεδρο Βεστάγερ δίνει ιδιαίτερη σημασία στο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και στην Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή εσείς είσαστε εκλεγμένοι και εκπροσωπείτε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, να σας ακούμε, γιατί με την πολιτική μας ανταγωνισμού προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολιτών μας. Πάντως θα έχετε διαπιστώσει, ελπίζω τουλάχιστον, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντάει σε κάθε ερώτηση που μας κάνετε χωρίς να χρησιμοποιούμε ξύλινη γλώσσα. Προσπαθούμε πραγματικά να απαντάμε στις ερωτήσεις σας γιατί ξέρουμε ότι αυτά που ρωτάτε είναι θέματα τα οποία απασχολούν ένα σωρό κόσμο. Οπότε σας διαβεβαιώνω ότι σε αυτήν την νέα επιτροπή Φοντερ Λάιεν με την Μάργαρετ Βεστάγερ αντιπρόεδρο η Επιτροπή και η αρμόδια επίτροπος θα συνεχίσει αυτόν τον καρποφόρο διάλογο μαζί σας. Τώρα θα έλεγα ότι μια από τις προτεραιότητές της και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς η ενίσχυση του ανταγωνισμού, της εφαρμογής δηλαδή των κανόνων ανταγωνισμού. Εγώ κάπου 30 χρόνια δουλεύω με τον ανταγωνισμό, πράγμα που δείχνει την ηλικία μου βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως είναι ο πρώτος χρόνος που έχει στο χαρτοφυλάκιο η Επίτροπος για τον ανταγωνισμό και εκείνη λέει ότι θέλει να πετύχουμε πολύ περισσότερα τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνεπώς, είμαστε προσανατολισμένοι ακριβώς στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Θέλουμε να εντοπίζονται τα προβλήματα, να επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης των περιπτώσεων αυτών και σε συνεργασία ε, μαζί σας να προχωράμε και με το δίκτυο επίσης που έχει δημιουργηθεί για τον ανταγωνισμό και όπου συμμετέχουν οι εθνικές αρχές. Προτεραιότητά μας είναι η αναθεώρηση πάντως κάποιων πτυχών των κανόνων ανταγωνισμού για το αντιτράστ, για τις συγχωνεύσεις και για τις κρατικές ενισχύσεις. Ακριβώς γιατί ξέρουμε τι γίνεται στις ψηφιακές αγορές, μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε μια παραδοσιακή, συντηρητική γενική διεύθυνση που θέλουμε να καθόμαστε και να κοιμάμαστε ήσυχοι χωρίς να ασχολούμαστε με τους κανόνες και την αναθεώρησή τους. Τώρα, για να είμαι σύντομος, γιατί θέλω να προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται περισσότερα σχόλια και ερωτήσεις σας, για τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Φυσικά υπάρχουν διεθνείς κανόνες και πρέπει να τηρούνται. Αυτό είναι ένας από τους κύριους πυλώνες μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα θα ήταν επιθυμητό ο ΠΟΕ να δρά, πώς να το πω, ε, πείθοντάς μας περισσότερο, με περισσότερο δυναμισμό. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία αλλά και οι Ηνωμένες συζητούν πώς τέτοιοι βελτιωμένοι κανόνες για τις επιδοτήσεις θα μπορούσαν ε, να, έχουν. Γίνονται διμερείς ε, συζητήσεις πάντως και με την Κίνα προκειμένου να πιστεί και εκείνη. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως, ως μέρος μιας ε, νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, ξέρετε ότι ο πρόεδρος Φοντερ Λάιεν ανέθεσε στην Επιτροπό μου, την κυρία Βεστάγερ, την ανάπτυξη μηχανισμών και πολιτικών για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι στρεβλωτικές επιπτώσεις επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία και ναι, γνωρίζουμε ότι κάποιοι από τους κύριους ανταγωνιστές μας παίζουν, πώς θα το πω, με διαφορετικούς κανόνες. Κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί με τα κατάλληλα μέτρα που θα υιοθετήσουμε. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση τώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την βελτίωση για να μην είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ για παράδειγμα, άλλους ανταγωνιστές ή να χρησιμοποιήσουν άλλους ανταγωνιστές. Φυσικά και αντιλαμβανόμαστε ότι διάφορες ε, ψηφιακές εταιρείε, δεν χρειάζεται να σας πω ονόματα τώρα, αγωνίζονται να έχουν ε, ολόκληρη την αγορά. Έχουμε μια ψηφιακή αγορά με επιχειρήσεις οι οποίες ακριβώς ε, επειδή υπάρχει αυτή η στρεβλή συμπεριφορά προσπαθούν να υποφεληθούν. Και γι' αυτό και γίνεται συζήτηση σε βάθος στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως μέσο διόρθωσης αυτού. Και εδώ άκουσα κάποιους από εσά να λένε ότι υψηλά πρόστιμα θα ήταν μια λύση. αλλά αποδεικνύεται ότι συχνά δεν ε, φτάνει. Γι' αυτό και προβληματιζόμαστε να δούμε μήπως θα έπρεπε να υπήρξε και κάτι άλλο από κατάσταση ας πούμε μέτρα, το οποίο όμως θα έπρεπε να δούμε ποια θα είναι για να δημιουργήσουμε ακριβώς ε, ισόρροπες συνθήκες ανταγωνισμού που πλήττεται βέβαια συχνά από τη συμπεριφορά αυτών των μεγάλων ε, ψηφιακών επιχειρήσεων. Τώρα δεν θέλω βέβαια να έχω παράσημα, αλλά να ξέρετε πάντως ότι ο αγώνας αντιτράστ που γίνεται για τις καταχρηστικές θέσεις κάποιων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο είναι κάτι το οποίο έχει στην πρώτη γραμμή και η Επίτροπος αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα θα γίνουν περισσότερα σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Αλλά αν ε, συγκρίνουμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, άλλες αρχές, άλλες χώρες, θα βγάλετε από μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Δεν είμαστε αφελείς. Μπορεί να είμαστε πολλά στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Αφελείς όμως δεν είμαστε. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ασφαλώς και γνωρίζουμε ότι κυρίως στις ψηφιακές αγορές ε, πολλοί υποστηρίζουν ότι η αγορά από μόνη της διορθώνεται και ότι δεν χρειάζεται παρέμβαση από τις δυνάμεις αντιτράστα, ε, αλλά βέβαια δεν ε, ισχύει αυτό, δηλαδή δεν σημαίνει ότι εμεί δεν θα κάνουμε τίποτα. Αλλά συγχρόνως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι θέλουμε να κάνουμε με τους κανόνες μας ανταγωνισμού. Εγώ και η Επίτροπος Φεστάκερ το έχει πει επανειλημμένος, οι κανόνες ανταγωνισμού, συγχώνευσης, αλλά γενικά οι κανόνες ανταγωνισμού, είτε είναι για τη συγχώνευση, είτε είναι για τις κρατικές επιδοτήσεις, αντιτράστη κτλ δεν πρέπει να εμποδίζουν την δημιουργία Ευρωπαίων πρωταθλητών. Όμως όπως κάποιοι από εσά το είπατε ήδη σήμερα το πρωί και συμφωνώ απόλυτα, η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτό το επιτυχάνουμε με αποτελεσματικό ανταγωνισμό πρώτα απ' όλα σε εμά μέσα στην Ευρώπη, γιατί μόνο έτσι οι δικοί μας πρωταθλητές μπορούν να δράσουν και να είναι πρωταθλητές και παγκοσμίως. Υπάρχει οικονομική ανάλυση και φαίνεται ότι αν δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο εσωτερικό, αυτό δεν είναι καθόλου καλή συνταγή για επιτυχία διεθνώς. Μπορούμε βέβαια, έρχονται για τα Χριστούγεννα, να είμαστε φιλόδοξοι και δεν πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε σε κακή κατάσταση οικονομικά ή όσον αφορά τη διεθνή μας παρουσία. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε ανοιχτή οικονομία με ανταγωνισμό, γι' αυτό και έχουμε σημαντικές επιχειρήσεις που δρούν και έχουν ηγετική θέση σε πολλούς κλάδους. Και τελειώνω. Αλλά εντάξει, εσείς με πιέσατε. Είπατε τόσα πολλά, τι να κάνω, να μην απαντήσω κι εγώ. Οπότε δώστε μου δύο λεπτά ακόμα, παρακαλώ. Όταν λοιπόν ε, μιλάμε για την χαλάρωση των κανόνων συγχώνευσης, προσοχή τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να γίνεται αλακάρτη η εφαρμογή των κανόνων, τότε δένεται τα χέρια της Επιτροπής σε διάφορους τομείς όπου υπάρχουν επιχειρήσεις απ' έξω που κυριαρχούν. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαφορετική προσέγγιση αν μια επιχείρηση είναι ευρωπαϊκή ή όχι. Τα PCI, όπως είπατε, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της ετοιμότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έχουμε γκρινει κονδύλια και το 2018 και το 2019 και θα έρθουν κι άλλα. Ναι, ακούω, βλέπω, μου λέτε πρέπει να σταματήσω. Τέσσερα λεπτά κανονικά έπρεπε να είχα. Το ξέρω, καταχράστηκα το χρόνο μου. Συγγνώμη να τελειώσω πάντως λέγοντας ότι η Επίτροπος Βαστέγερ σκοπεύει να κρατήσει ανοιχτές αυτές τις συζητήσεις και μαζί σας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Η εχει έχει δύο-τρία λόγια για τα καταληκτικά της σχόλια. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω λιγότερο από 10 λεπτά που μίλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι παρόλα αυτά που βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ επικοδομητικά σας σχόλια που προλέγουν θα γίνουν πάρα πολύ καλές ανταλλαγές απόψεων. Ε, βλέπω ότι ακόμα και εσωτερικά πολλών πολιτικών ομάδων υπάρχουν διστάμενε απόψει, γιατί αυτό, και αυτό είναι καλό και θα εμπλουτίσει το κείμενό μα. Έχω τρία γενικά σχόλια. Πρώτον, όπω ξέρετε, καλύτερα από μένα, γιατί είμαι καινούρια Ευρωβουλευτή, είναι πολύ απογοητευτικό να φτιάξει κανεί μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τελικά ε, έχουμε 6.000 ε, στοιχεία μόνο. Χαρακτήρε. Εστρέφομαι εδώ προς την γραμματεία ε, γιατί μου επέβαλε αυτό το όριο και τελικά έφτασα στο 5.999 ας πούμε. Είχα πολλά να πω. Ε, βλέπω ότι θα τα προσθέσετε αυτά τα που δεν είπα εγώ, εσείς εν είδη τροπολογιών. Πρέπει να βρούμε κάποια ισορροπία ανάμεσα στη, στα γενικόλογα σχόλια και στα πολύ πολύ εξειδικευμένα. Ε, νομίζω ότι οι τροπολογίες θα μας βοηθήσουν να συγκεκριμενοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι ε, όταν μας επιβάλλονται τους περιορισμούς 6.000 χαρακτήρων, ε, είναι λίγο απογοητευτικό. Τώρα, για τον κύριο Έπινγκ, να απαντήσω. Επιβεβαιώνω ότι υπέβαλα το σχέδιο έκθεσης ε, τη μέρα που μπήκε και στο διαδίκτυο. Σχέδιο έκθεσης, προσχέδιο μάλλον έκθεσης. Ε, κύριε Έπινγκ, υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο, γιατί είμαι καινούργια όπως σας είπα. Ε, αν έχετε αντίρρηση, ας πούμε, ε, αν υπάρχει κανόνας που μου απαγορεύει να κάνω κάτι τέτοιο, ε, να το ξέρω. Μέχρι να υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια, είναι σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Και επομένω τίποτα δεν με απαγορεύει, μια και δημοσιεύτηκε ούτω ή άλλω ε, σε γαλλική γλώσσα στα στο διαδίκτυο, εξάλλου η κυρία Βεστάγκερ ε, μιλάει και καλά γαλλικά, μου φάνηκε ότι ενδιαφέρον να της το δώσω τη μέρα που ούτως ή άλλως δημοσιευόταν ε, στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν έκανα κάποια παράβαση, κάποιο λάθος, να μου το πείτε. Θα ήθελα να το ξέρω για την επόμενη φορά, γιατί την πρώτη μου έκθεση. Ε, δείξτε λίγη κατανόηση και ανοχή. Έσφαλα καλόπιστα. Τώρα για την πρακτική της ε, κατηγορίας ε, στηλίτευσης εταιριών. Δίστανται οι απόψεις. Εγώ νομίζω ότι στις ε, προηγούμενες εκθέσεις το κάναμε αυτό συστηματικά. Ε, οι υποθέσεις που αναφέρονται είναι πασίγνωσες υποθέσεις. Ε, τα ΜΜΕ μίλησαν πάρα πολύ για αυτές. Είναι εμβληματικέ υποθέσεις. και όλοι συμφωνούμε μια και εκπροσωπούμε όλοι πάνω από 510 εκατομμύρια ε, πολιτών και καταναλωτών, ε, κάπως θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Γιατί να αφήσουμε μόνο τα ΜΜΕ να κάνουν αυτό το ρόλο. Θα πρέπει και εμείς να παίξουμε το δικό μας παιδαγωγικό ρόλο. Βεβαίως, η λέξη στυλίτευση είναι λίγο αρνητική, έχει αρνητική χρειά. Δεν θέλω να κατηγορήσω αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιχειρήσεις τις οποίες, ε, στις οποίες επιβάλλουμε κυρώσεις, θέλω απλώς να αναφέρω κάποια στοιχεία. Για παιδαγωγικούς λόγους πάντα. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της, για τα ενδιαφέροντα της σχόλια που προλέγουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ Κάρμεν για το ραντεβού σε λίγους μήνες, ούτως ώστε να δοθεί συνέχεια και, την, ε, και να πουλήσουμε καλά αυτή την ε, έκθεση. Και μάλιστα και μετά τη δημοσίευσή τη να συνεχίσουμε να την διαφημίζουμε. Ε, τώρα, για την έκθεση αυτή έχετε προθεσμία ε, μέχρι τον Ιανουάριο 9 για τροπολογιε 22 22-23 θα τι εξετάσουμε τις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και εν συνεχεία θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Και με αυτά περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση για, τις, για τους διαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων. Είμαι η συγγήτρια μαζί με την Εστέρ Ντε από το, ΕΛΚΑ. Η Έστερ έχει το λόγο για να παρουσιάσει την έκθεση. Οκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Συνεισηγήτρια για όσοι είστε νέοι, το θέμα αυτό το κληρονομήσαμε από την προηγούμενη θητεία κατά κάποιο τρόπο. Τότε ήμουν συνεισηγήτρια με τον προκάτοχό σας, τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, κυρία Πρόεδρε. Και ήδη είχαμε καταλήξει σε μια κοινή θέση δύο συνεισηγητές. Μπορεί να είναι τεχνική αυτή η έκθεση, αλλά είναι και ευαίσθητη και λεπτή. Εμείς οι δύο τώρα ως ναι εισηγήτρες. Εσείς είστε νέα, εγώ είμαι παμπάλαια. Αλλά ε, αποφασίσαμε να καταθέσουμε την ίδια έκθεση που είχα κάνει με τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Μπορεί να θυμάστε ε, ότι στο θέμα των κόκκινων δανείων στα μη εξυπηρετούμενα Συμφωνήσαμε ε, για την προληπτική προστασία, prudential backstop, για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις για τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, εδώ μιλάμε ε, για μια νέα οδηγία και για να την περιπλέξουμε περισσότερο την έχουμε σπάσει στα δύο και τώρα συζητάμε σήμερα το πρώτο τμήμα που έχει να κάνει με τις δευτερογενείς αγορές. Αυτή η οδηγία φυσικά έχει επιπτώσεις και για τα κράτη-μέλη και για τους καταναλωτές και άλλους φορείς της αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό να τα ρυθμίσουμε σωστά αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν κάποιες αρχές που μας καθοδηγούσαν από την αρχή, περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία ε, για να μπορούν τα κρατη να αντιμετωπίσουν αυτό το υψηλό όγκο κόκκινων δανείων, προστασία των ε, καταναλωτών και των μικρομεσαίων δανείων λιπτών, να μην καταργήσουμε την ένωμη τάξη των κρατών μελών και συνεργασία για το ξέπλυμα ε, και τις ασφαλιστικές δικλείδες. Και χαίρομαι που μείναμε σε αυτές τις αρχές. Μπορεί να υπάρχουν κάποια ε, θέματα που θέλετε να σας αναφέρω για το περιεχόμενο. Το πεδίο εφαρμογής είναι πολύ στοχευμένη η έκθεσή μας, ειδικά για, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τις, ε, ε, ε, την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Έχω επικεντρωθεί εκεί. Δεν θέλω να σας δώσω το πλήρη κατάλογο. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν σημασία για τους συναδέλφους. οι ε, όροι δανειοδότησης δεν μπορούν να αλλάζουν μόνο μερός. Αυτό έχει να κάνει με την προστασία των καταναλωτών. Ε, θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά οι δανειολήπτες, τα λεφτά του άρθρου 13. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ενημερώνουν καλύτερα αν θέλουν. Υπάρχει μια μήνυμο με εναρμόνιση, αλλά αν θέλουν περισσότερη πληροφόρηση μπορούν να το κάνουν. Όπως είχα πει και στην περασμένη θητεία ε, για την εξοδικαστική διαδικασία την επιταχυμένη ε, στο μεταξύ, μιλώ τώρα εξ ονόματος μου μόνο, το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε κοινή θέση για το δεύτερο τμήμα της οδηγίας, μάλλον και για το δεύτερο, και προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε κινήσει και στο δεύτερο τμήμα αυτή τη οδηγίας. Όπω γνωρίζετε όλο αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων συνδέεται και με άλλε συζητήσει που έχουμε για την Τραπεζική Ένωση και καλό θα ήταν να δείξουμε ότι προχωρούμε και κινούμαστε σε αυτό το θέμα για να προχωρήσει η υπόθεση τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάντως που με αφήσατε να σας περιγράψω κάποια. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε και περιμένω να ακούσω ε, τις απόψεις των συναδέλφων. Στο Μέστερ, είπε ήδη κάποια από τα βασικά θέματα. Θα ήθελα λιγάκι να πάω προς τα πίσω, να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω και να υπενθυμίσω το συνολικό πλαίσιο και τη σημασία αυτού του κειμένου, που είναι στοιχείο ενός, μιας κλήρου στρατηγικής που αποφασίζει το Συμβούλιο για τη μείωση του όγκου το μη εξυπηρετούμενο δανείο, τον αποφάσισε τον Ιούλιο του 2017, για να ενισχύσει ε, την προληπτική εποπτεία ε, με τον προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας. Θα πρέπει να έχουμε μια ε, λειτουργική δευτερογενή αγορά για τα προβληματικά δάνεια. Είναι πρόβλημα που οι συνομοθέτες έχουν ήδη αντιμετωπίσει ε, με τον κανονισμό Μίξ Πρετούν δανείων, όπου έχουμε καλύτερε διατάξεις για τα πιστοτικά ιδρύματα, τα οποία αγοράζουν τέτοια δάνεια. Ε, το μέλημά μα ήταν διτό, ε, από τη μία να βοηθήσουμε μία εύρυθμη δευτερογενή αγορά και να έχουμε και ένα σαφές νομικό πλαίσιο για αυτή την αγορά, με σαφείς κανόνες εποπτείας για τους αγοραστές και την κατάλληλη προστασία για τους δανειολήπτες. Ε, είχαμε τις ίδιες ανησυχίες με αυτές που ανέφερε η Έστερ, ε, συντάσσοντας αυτήν την έκθεση. Συμφωνούμε με το βασικό στόχο της Κομισιόν. Ε, η πρόταση της Κομισιόν όμως έχει δύο ελλείψεις. Καταρχάς, δεν λαμβάνει σωστά υπόψη το γεγονό ότι οι κανόνε για την αγορά πιστώσεων και τη διαχείριση των πιστώσεων αυτή τη στιγμή διαφέρουν πάρα πολύ από κράτο σε κράτος. Ε, έχουμε πολύ φιλελεύθερε προσεγγίσεις από τη μία άκρη του σε πιο ε, περιοριστικές. Και επομένως ε, μια μεγαλύτερη εναρμόνιση και το διαβατήριο για τι πιστοτικέ υπηρεσίε ε, σε όλη την Ευρώπη θα ήταν κάτι θετικό. Το να προτείνουμε εναρμόνιση με ελάχιστε απαιτήσει μόνο δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Στη γενική προσέγγιση, το Συμβούλιο κράτησε τι ελάχιστε ε, προποθέσει αυτέ και έβαλε τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη, αν θέλουν, να ζητήσουν επιστοτικέ ε, υπηρεσίε να αυτές να πληρούν ε, πιο αυστηρές προϋποθέσεις, υποσκάπτοντας, α πούμε, το στόχο της εναρμόνισης που είναι ο στόχος της οδηγίας. Στο σχέδιο έκθεσης, λοιπόν, έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή να έχουμε πιο αυστηρές απαιτήσει που θα εφαρμόζονται παντού. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων ε, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίσουμε επαρκή ε, χρηματοδότηση και προϋποθέσεις ε, ε ρευστότητας, ε, σωστή διαχείριση, προστασία, προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρουσία κανόν, σωστών κανόνων για να διαχειρίσουμε και να μετριάσουμε τον κίνδυνο. Οι πιστοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν επαρκείς διαδικασίε κάτω του ξεπλήματο του χρήματος, η δεύτερη έλλειψη της πρότασης Κομισιόν είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη κάποιες αφέλτες ε, επιπτώσεις. Το σκοπό της ανάπτυξης της δευτερογερνούς αγοράς για όλα τραπεζικά δάνεια που μπορεί να ευνοήσει ε, κάποια επιχειρηματικά μοντέλα σε κάποιες περιφέρειες όπου οι τράπεζες δεν ε, ελέγχουν σωστά την αξιοπιστία κάποιων δανειοληπτών και μεταβιβάζουν αυτέ τι πιστώσει εύκολα. Και αυτό μπορεί να υποσκάψει την προστασία των δανειοληπτών. Γι' αυτό το σχέδιο, στο σχέδιο έκθεση αποφασίσαμε να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή εφαρμογή, εφαρμογής οδηγία μόνο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίση, για να εξασφαλίσουμε ε, προστασία των οφειλετών και να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα των δευτερογενών αγορών, οι αγοραστές ε, πιστώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις, ε, τους εποπτικούς φορείς των πιστοτικών ας πούμε, ιδρυμάτων για τη διαχείριση των πιστώσεων που αγοράζουν, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και, την, και το είδος του οφειλέτη. Αυτό θα προστατεύσει όχι μόνο τον καταναλωτή, αλλά όλους τους δανειολήπτες και τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Μια η εποπτεία ε, Μπορεί να μην είναι πολύ σωστή, θα θέλαμε οι πιστοτικέ υπηρεσίες που ε, να είναι οντότητε που εποπτεύουμε γενικά. Επανέρχομαι σε αυτό που αρχικά. Να δημιουργήσουμε μια πραγματική ε, πανευρωπαϊκή δευτερογενή αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δράνεια για να έχουμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας καταναλωτών και ε, δανειοληπτών. Αυτά είπαμε στην εκθεσή μας. Αυτά είναι τρία βασικά στοιχεία. Δεν θα αμφισβητηθούν ούτε στην τελική έκθεση, ούτε στη μελλοντική πιθανή συμφωνία με το Συμβούλιο, γιατί είναι τρεις πυλώνες ε, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντίθετα από τις αριστολογίες εδώ πέρα ε, των Βρυξελών. Υπάρχουν ε, αρμοδιότητες που έχουν οι εθνικές αρχές, ε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε παντού ευρωπαϊκή διάσταση, ε, έστω ας πετύχουμε αυτή την νομοθεσία, αυτό να μην έχουμε καμία νομοθεσία για αυτό το θέμα. Αυτό είναι καλύτερο για τους πολίτες. Είμαι έτοιμη να ακούσω τα σχόλιά σας. Ξεκινάμε τους κοιόδης εισηγητές. κύριος Αγγίν από το Renew. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πλευρά τη ομάδα Renew είναι πολύ καλό το σχέδιο έκθεση. Εγώ είμαι και ο και ασχολούμαι με αυτή. Κατά την άποψή μα αποτελεί καλή βάση, εξαιρετική βάση εργασία για να δούμε τα προβλήματα των κοκκίνων δανείων και των τραπεζών. Θα πρέπει ε, σίγουρα να κάνουμε τροπολογίες ε, από το Ρινιού. Ήδη το γραφείο μου έχει αρχίσει να τις γράφει. Είναι πολλά τα καλά, αλλά υπάρχουν και μερικά θέματα που μας ε, έκαναν εντύπωση. σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ε, πρακτικό. Η γραφειοκρατία στην πώληση των κόκκινων δανείων παραμένει ψηλή. Μέχρι να πουλήσει αυτό το δάνειο μία τράπεζα, φτύνει αίμα. Ειδικά όταν έχει πάρα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Χρειάζεται να προσλαμβάνει προσωπικό για να πουλήσει τα δάνεια. Χρειάζονται μηχανισμοί ε, που να το αντιμετωπίζουν αυτό. Είναι καλή έκθεση και ισορροπημένη, αλλά πρέπει να προτείνουμε τέτοιες λύσεις και χαίρομαι για την επικοδομητική συνεργασία που σίγουρα θα έχουμε. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Προχωρούμε ο κύριο Σουρτάσον είχε ένα οικογενειακό θέμα. Δεν ξέρω ποιο είναι από τους πρασίνους εδώ επίγον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα σας διαβάσω αυτά που μου έδωσε ο κύριο Σουρτάσον. Λέει ο κύριο Γιακελιούνα. Ε, ε, τα είχε γράψει πριν ακούσει αυτά που είπατε εσεί οι δύο εισηγήτριε. Στο τέλος θα σας δώσω και την προσωπική μου άποψη, πολύ ε, σύντομα. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τι ε, συνεισηγήτριε για το σχέδιο έκθεση που αντανακλά τη θέση τη προηγούμενη έκθεση περασμένη θητείας. Είναι ρητό ο στόχος ε, την πρόταση της Οδηγίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών για να μπορούν οι τράπεζε να πολλούν τα κακά δάνεια και να τα διαχειρίζονται. Αυτό που λείπει και μα κάνει εντύπωση από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελείω από την αιτιολογική έκθεση και τη μελέτη αντικτύπου είναι η προστασία των καταναλωτών όπου το πρόβλημα των κόκκινων δανείων οφείλονται κυρίως στην ανευθυνότητα ε, της πολιτικής χορηγήσεων των τραπεζών. Και δεν φταίνε οι καταναλωτές, αλλά τους έχουν κατακλείσει οι τράπεζες με κακά δάνεια. Ε, σε αντίθεση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δύο συνεισηγήτριες βάλατε επιπλέον κριτήρια για την έγκριση των ε, χορηγήσεων αυτών για καλύτερη ρύθμιση ε, αυτών των ε, καταστάσεων. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να υπερψηφίσουμε στην ε, περασμένη θητεία του συμβιβασμούς και παραμένουν οι επιφυλάξεις μας για να υπάρχει επαρκής προστασία των καταναλωτών. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τις επιστοτικές υπηρεσίες, αλλά και όλο αυτό το εμπόριο το δευτερογενές που γίνεται με τα δάνεια. Και αυτό θα πρέπει να το δούνε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συγγήτρες, γιατί δεν προτείνουν τίποτα σχετικά. Επίσης, θέλουμε να δούμε στο κείμενο και στις διαπραγματεύσεις ε, κάποια μέτρα σχετικά με την υποχρέωση των πιστωτών και θα κάνουμε τέτοιες τροπολογίες ε, για ενημέρωση στο δανειολήπτη όταν ε, υπάρχουν νέοι ευνοϊκοί για εκείνον όροι ε, και αναδιατύπωση της δανειακής σύμβασης. Θα κάνουμε σχετικές τροπολογίες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις διάφορες τις πρακτικές εταιρείες και τις πρακτικές που ακολουθούν και τη συμπεριφορά τους θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πολύ καλά ποια κριτήρια ισχύουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην έχουμε καταχραστικές ε, καταχρηστικές πρακτικές όπως βλέπουμε από διάφορες πρακτικές εταιρείες σε πολλά κράτη-μέλη. Επίσης, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενημερώνονται με σωστό τρόπο και αυτό θα πρέπει ε, να γίνεται με τεχνικές ε, προδιαγραφές υποχρεωτικές για τις τράπεζες και όχι με κάποια εθελοντική ε, πρόταση. Η οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί ε, στην Εθνική Ένωμη Τάξη κάθε φορά με μεγάλη ευελιξία, αλλά να μην είναι γενικόλογες οι υποχρεώσεις και σε επίπεδο διακηρυκτικό μόνο, αλλά δεσμευτικές αυτές που πρέπει να αναλαμβάνουν. Το Μητρό στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, που προτείνεται είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς να απελευθερώσουμε όλες τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να αυξηθούν ε, τα στάνταρ προστασίας των καταναλωτών. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μας. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ε, επίφοβα αυτά τα δάνεια, είναι μεγάλα τα ποσά, είναι μεγάλα και τα χρονικά διαστήματα αποπληρωμής και μπορεί να συμβούν διάφορα πρόπτα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν οι δανειολήπτες. Και το θέμα της εποπτείας είναι και αυτό σημαντικό. Τα στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να τα δούμε ειδικά, ξεχωριστά, γιατί είναι πολλά σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρκο Τζάνι από την ομάδα ID. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τις δύο συνεισηγήτριες για τις προτάσεις τους, οι οποίες πιστεύω ότι ε, πολύ θετικά βελτιώνουν κάποιες από τις επικρίσεις που είχε η Επιτροπή. Και χαίρομαι που μιλάτε για περισσότερη διαφάνεια και κυρίως που μιλάτε για σωστές διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητας ή κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τώρα, στις συζητήσεις που θα έχουμε με τις συζητήτριες και τους σκιώδες συζητητές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε ένα καλό πλαίσιο. Πρέπει να δουλέψουμε για την διαφάνεια, αυτή είναι η πρώτη αρχή και με την οποία όλοι συμφωνούμε νομίζω, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτού του είδους ε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και στα πλαίσια που δρούν οι διάφορες αγορές, η διαφάνεια είναι κάτι δύσκολο. Οπότε θα βοηθήσει πολύ και τις δευτερογενείς αγορές. Άρα να δουλέψουμε πάνω στη διαφάνεια. Το δεύτερο θέμα που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι η προστασία των καταναλωτών που πρέπει να αποτελέσει μια κατευθυντήρια γραμμή προς όφελος των δευτερογενών αγορών. όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ποιος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ποιος δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάποια τέτοια οδηγία. Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής δεν το κάνει ακριβώς και νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν και ισόρροποι κανόνες, ίδιοι για όλους. Ισότιμοι, αν με τι άλλο. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά και οι προτάσεις από τις συνεισηγήτριες πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω εδώ. Και θα τελειώσω με μια γενική πολιτική παρατήρηση που έχει να κάνει και με την πρόταση της Επιτροπής. Δηλαδή, προσοχή να μην στενέψουμε πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογής και μην επιβάλλουμε υπερβολικό άχθος πάνω στον τραπεζικό κλάδο. Έχει γίνει ήδη πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά τα μη ξυπηρετούμενα δάνεια. Και ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν έχει επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τις αγορές να το κάνουμε. Να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν είναι και ο μόνος κίνδυνος που ελοχεύει στους ισολογισμούς των τραπεζών. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε υπερβολικά σε αυτό και δώσουμε ιδιαίτερη σε αυτό το ζήτημα, ε, τότε φοβάμαι ότι θα χάσουμε το στόχο της οδηγίας που είναι να δημιουργήσει αποτελεσματικές δευτερογενείς αγορές και κινδυνεύει να κάνει περισσότερη ζημιά από ότι να λύσει τα υπάρχοντα προβλήματα. πάντω, θα δουλέψουμε και εμεί πάνω σε τροπολογίε και προβλέπουμε στις συζητήσει. Ευχαριστώ. Κύριο Σέπι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση της κυρίας Ντελάνκε και η δική σας είναι μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουμε και χαιρόμαστε ε, για όσα αναφέρονται όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή ε, να υπάρξει παρέμβαση από εξωτερικές ε, επιχειρήσεις και για όλα τα δάνεια, επειδή η ελεύθερη αγορά μπορεί να φροντίσει. Έπειτα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, έχουμε ήδη νομοθεσία που το καλύπτει. Προσβλέπουμε λοιπόν σε επικοδομητική συνεργασία και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδημούλης τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριες ε, για τις προτάσεις τους. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός <clears throat> ο τρόπος με τον οποίο θα επιμεριστεί ο κίνδυνος για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια <clears throat> στον ιδιωτικό τομέα μέσω της δημιουργίας μιας δευτερογενούς αγοράς για την πολιτική μου ομάδα και για μένα προσωπικά ε, αποτελεί προτεραιότητα αυτή η διαδικασία να εξασφαλίζει την πληρέστερη δυνατή προστασία στους πιο αδύναμους δανειολήπτες καταναλωτές, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν στεγαστικά δάνεια και σε αυτούς που το στεγαστικό δάνειο αφορά την πρώτη τους κατοικία. Πρέπει η προσπάθεια δηλαδή να μην επιδιώκει με τη θέσπιση των κανόνων να βοηθήσει απλώς τις τράπεζες να βελτιώσουν τα λογιστικά τους βιβλία, αλλά να παρέχει και την προστασία που απορρέει από το άρθρο 7 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δανειολήπτες πρώτης κατοικίας και στους καταναλωτές. Γι' αυτό υπάρχει μια ανάγκη οι κανόνες να είναι πολύ αυστηροί και όσον αφορά την αξιοπιστία και τον έλεγχο των εταιριών που ασχολούνται στη δευτερογενή αγορά ακινήτων με αυτά τα θέματα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε εκεί μια πειρατική δραστηριότητα. Χρειάζεται να έχουν νομική υπόσταση, να έχουν αδειοδότηση από τα κράτη-μέλη. Δεν είμαστε καθόλου σύμφωνοι να μπορεί μια εταιρεία να έχει έδρα σε μια χώρα και να έχει ένα ιονί διαβατήριο για να λειτουργεί και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Όπως επίσης πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο ανοιχτοί όσο η πρόταση η αρχική σε θυγατρικές πιστοτικών ιδρυμάτων καθώς δεν είναι όλες οι θυγατρικές εποπτεγόμενες από τις χρηματοπιστωτικές αρχές. Με αυτό το πνεύμα που λέει ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε την αναγκαστική εκτέλεση ε, σε ό,τι αφορά δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και κοινωνικά ευαίσθητοι στους αδύναμους καταναλωτές δανειολήπτες και ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, θα καταθέσουμε προτάσεις, τροπολογίες προς τις δύο συνεισηγήτριες ε, και ε, προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία έτσι ώστε να επηρεάσουμε το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα επικοδομητικά σας σχόλια και τις προτάσεις σας και τη διαθεσιμότητά σας για συνεργασία. Δεν έχεις στήσει κανείς το λόγο στο Κατσδιά. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην Έστερ, νομίζω, για να απαντήσει. Όχι, μόνο να ευχαριστώ αδέρφους θέλω για το όσα είπαν. Κάποιοι από εσά ήδη είπατε ότι θα φροντίσετε και συμβαστικές τροπολογίες. Ωραία, θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να πετύχουμε ευρεία πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης αυτής. Το μόνο που μένει τώρα είναι να θυμίσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αλλά αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Πρόεδρος, ναι. Ωραία. Κλείνοντας, να κάνω κάποια σχόλια για την ανάγκη για επιπλέον απαιτήσει. Κάποιες τράπεζες ήδη έχουν τέτοιες απαιτήσει που πρέπει να σέβονται και να τηρούν. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγέ, ενίσχυση, επανενίσχυσή τους, αλλά προσέχοντας βέβαια να μην δημιουργούμε επικαλύψει. Να ξέρουμε τι ήδη υπάρχει και τι θέλουμε να πετύχουμε. Οι άλλες ανησυχίες για την διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών, Βεβαίω είναι και οι δικές μας κύριες ανησυχίες. Όσο διαμορφωνόταν η έκθεση αυτή και από τους προκατόχους μας και από μας. Φυσικά και θα ανταλάβουμε υπόψη μας αυτά. Όσον αφορά την αποσταθεροποίηση του συστήματος, εάν επιμείνουμε υπερβολικά στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτό το είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία, ε, όλα αυτά να πηγαίνουν χέρι-χέρι με την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εννοείται ότι αυτή είναι η ανησυχία μας και ότι θέλουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι σταθερά. Είναι προς το συμφέρον όχι μόνο του κλάδου, αλλά και προς το συμφέρον των καταναλωτών και των πολιτών. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 19η του μηνός στις 2 το μεσημέρι. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 27 και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 17-18 Φεβρουαρίου. Στην Ολομέλεια πότε θα πάει, τον Μάρτιο? Ωραία, τελειώσαμε για σήμερα. Οι επόμενες συνεδριάσεις μας είναι 13 Ιανουαρίου, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και μετά, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, 9 με 12.30 και 2.30 με 6.30 και την 5η 23 Ιανουαρίου, 9 με 12.30. Ευχαριστώ πολύ.